Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κηρύξω την έναρξη της απογευματινής μας συνεδρίασης. Όπως γνωρίζετε, σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό προσκεκλημένο, προσκεκλημένη για την ακρίβεια, Όλα καλά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω την ξεχωριστή μας καλεσμένη, την οποία συνοδεύει και μέλης αντιπροσωπεία. Θα ήθελα να της εκφράσω την ικανοποίησή μου και τη χαρά μου που μπόρεσε να έρθει μαζί με την αντιπροσωπεία με μέλη της κυβέρνησης Βραζιλίας και της Βουλής της Βραζιλίας. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας γιατί γνωρίζουμε τα σημαντικά επιτεύγματα και τους ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης της βραζιλιάνικης οικονομίας. Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις σχέσεις της Βραζιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και να σας καλωσορίσω θερμότατα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, κυρία Αμπρέου. Όπως είπα, σε συνοδεύει πολυμελής αντιπροσωπεία από βουλευτές και γερουσιαστές. Ο Ιερουσίας της Ρέμος, για παράδειγμα. Αναστάζια. Ο Ιερουσίας της Μάρτινς. Φίλιο Λαμπρέου. Ο κύριος Καλέπκο. του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού και ο κύριος Κομπίνεν και φυσικά και ο πρέσβης ε, της Βραζιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Μασάντο. Δεν μπορώ να αναφέρω ε, ξεχωριστά όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας. Σας καλωσορίζω πάντως θερμά. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας ε, για τη σχέση με τη Βραζιλία, την κυρία Ζαλίνο. Καλώς ήρθατε. Όπως είπα και προηγουμένως, η, η Υπουργός εξέφρασε την επιθυμία στη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συναντηθεί με την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Γεωργίας, γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις μας, ε, οι εμπορικές, με τη Βραζιλία γιατί είναι σημαντική η γεωργία, η κτηνοτροφία στη Βραζιλία και μεγάλος όγκος των βραζιλιάνικων ε, εξαγωγών. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Σας ε, καλωσορίζω θερμότατα για μια ακόμη φορά και σας δίνω κυρία Υπουργέ το λόγο. Μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια στους λοιπούς βουλευτές για να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και τις απορίες τους. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ας μην καθυστερούμε άλλο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Γεωργίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σεκέρσκι. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και να χαιρετήσω θερμότατα όλα τα μέλη αυτής της πολύ σημαντικής επιτροπής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Βραζιλία. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους τεχνικούς συμβούλους, τους υπαλλήλους, τους δημοσιογράφους και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι με συνοδεύει η αντιπροσωπεία βουλευτών από τη Βραζιλία. Ήδη πήγαμε στο Παρίσι, στι εντρίες του ΙΕ, σήμερα είμαστε στις Βρυξέλλες και θα πάμε μέχρι τη Γενέβη. Ε, η Άννα Μέλια Λέονς είναι από την ε, Βρασιλιανική Γερουσία και είναι και πρόεδρος της ε, Επιτροπής Γεωργίας στη Γερουσία, στην Ομοσπονδιακή Γερουσία. Και ο κύριος Αβραίου είναι πρόεδρος Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής. Ο γερουσιαστής Μαρτίν από το Ρίο Γκράντε του Σούλ, ο γερουσιαστής Αντώνιο Αναστασία από την πολιτεία Μίνα Ζεράης, πρώην κυβερνήτης ε, ε, μιας πολύ σημαντικής πολιτείας της Βραζιλίας ε, και είναι της, ο βουλευτής Βα... Βαουτζίρ Κολάντου από την πολιτεία της Σάντα Καταρίνα, ο κύριος Κροβινέολ, βουλευτής από την Κογιάς, από την περιφέρεια Κογιάς και θα ήθελα να, να ευχαριστήσω θερμά την πρέσβη Βέρα Μαρτίνς για τη θερμή υποδοχή στις Βρυξέλλες και φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπής και τους τεχνικούς που μας συνοδεύουν. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητά και αξιότιμα μέλη, ε, εξοχότητες, ε, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να απευθύνω ομιλία στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα να το κάνω ως Υπουργό Γεωργίας της Βραζιλίας. Θα ήθελα να σας εξηγήσω με λίγα λόγια τα οράματα της πατρίδας μου σε ό,τι αφορά την παραγωγή και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων καθώς και το θέμα της προσφοράς τροφίμων για όλο τον πληθυσμό του πλανήτη γιατί όσο θεμητά και αν είναι τα ιδιαίτερα συμφέροντα της κάθε χώρας, τα θέματα της γεωργίας και της διατροφής είναι ακόμη πιο σημαντικά και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ικανή παραγωγή αγροτικών προϊόντων για την ικανοποίηση των αναγκών όλου όκληρου του πληθυσμού της γης, ώστε να έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες χωρίς εξαίρεση. Και παρά τις διακοιμάσεις που είχαμε στην ανάπτυξη στις πλούσιες χώρες τα τελευταία χρόνια, ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες, διαπιστώσαμε ότι υπήρξε τεράστια και γενικευμένη ε, πρόοδο σε ό,τι αφορά τη μείωση της ε, ακραία φτώχεια, τη εξαθλίωση σε όλα τα πάρη του κόσμου. Και ε, τώρα τελευταία είχαμε πραγματικά μια άνευ προηγουμένου πρόοδο, γιατί εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, ιδιαίτερα στην Ασία και την Λατινική Αμερική, ε, ξεπέρασαν την εξαθλίωση και την ακραία φτώχεια και μπόρεσαν ε, να μπουν στον κόσμο της κατανάλωσης και της επίσημης εργασίας. Και αυτή η πολύ θετική αλλαγή που είναι ευπρόσδεκτη για όλους, ε, συνιστά και μια τεράστια πρόκληση για την γεωργική παραγωγή. Στις περισσότερες χώρες η χρήση της γης για την γεωργία και την κτηνοτροφία έχει φτάσει στα ωριά του. Και μόνο εξαιρετικά η αύξηση της παραγωγικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής εντυπωσιακή. Ταυτόχρονα οι πληθυσμοί θα ο πληθυσμός θα, να, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Όλοι γνωρίζουμε ότι γύρω στο 2050 θα έχουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια επιπλέον ε, κατοίκους και καταναλωτές. Οπότε έχουμε και διοντολογικές ανάγκες και ηθικές και πρακτικές. Θα πρέπει να παράγουμε περισσότερα και καλύτερα πιο ποιοτικά τρόφιμα που θα είναι προσιτά σε όλους. Γιατί αν δεν σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και δεν εξασφαλίσουμε παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε πολιτική και κοινωνική αστάθεια στις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου. Ε, και μάλιστα με συνέπειες που μπορεί να γενικευθούν και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Βραζιλία μαζί με κάποιες άλλες χώρες ε, μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στην ε, πολύ αυτή σημαντική διάδοση και εξάπλωση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Εμείς έχουμε 8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Μόνο όμως 28% της έκτασης αυτής χρησιμοποιούνται για την γεωργία και την κτηνοτροφία και ανήκουν ε, σε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Ε, γιατί αν ε, διακρίνουμε το, αυτό από το 11% των πόλων και των ε, υδάτινων λεγάων, έχουμε μόνο 61% στη Βραζιλία, 61% της επικράτειάς μας, που αποτελούν προστατευμένες ε, οικολογικές περιοχές. Και χάρη στους κώδικες που έχουμε και τους περιβαλλοντικούς ε, νόμους μας, που είναι από τους πιο αυστηρούς ε, και διεξοδικούς του κόσμου, έχουμε ακόμη ένα, μια τεράστια έκταση για να διαβρύνουμε την παραγωγή μας. είτε ε, περιλαμβάνοντας νέες περιοχές ε, όπως επιτρέπουν οι κανόνες ή ανακτώντας ε, την παραγωγικότητα σε περιοχές που δεν έχουν μεγάλη παραγωγικότητα ή αναβαθμίζοντας ε, κάποιους βοσκοτόπους. Από το 2002 μέχρι σήμερα, μεταξύ των μεγάλων παραγωγών γεωργικών προϊόντων του κόσμου, όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες, η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδία και η Ρωσία, η Βραζιλία ήταν η χώρα που είχε τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας. Από το 1970 όταν ξεκίνησε η γεωργική μας επανάσταση, είχαμε σταθερά αυξήσεις της παραγωγικότητας. Και τα τελευταία 20 χρόνια η αύξηση της παραγωγικότητας της γης μας μας επέτρεψε να εξοικονομήσουμε περίπου 50 εκατομμύρια μονάδες ε, μόνο στην παραγωγή δημητριακών. Έχουμε ε, εδάφη λοιπόν, γεωργούς και τεχνολογίες εχμής, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας, κυρίως μέσω της αύξησης παραγωγικότητάς μας. Και οι μελέτε και οι προσωμιώσει μα λένε ότι με δεδομένε και τι ίδιε οικονομικέ συνθήκε θα μπορέσουμε την επόμενη δεκαετία να αυξήσουμε ε, κατά 50 εκατομμύρια τόνους την παραγωγή δημητριακών και 8 εκατομμύρια, κατά 8 εκατομμύρια τόνους ε, την παραγωγή βοηού κρέατος, χείριου και πουλερικών, χωρίς αυξήση, αύξηση της αποψήλωσης. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η βραζιλιάνικη παραγωγή είναι διεθνώς ανταγωνιστική για εύλογους λόγους. Έχουμε αυστηρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους που εξασφαλίζουν όχι μόνο τη διαφύλαξη του, της περιοχής του Αμαζονίου και της οικολογικής ζώνης αυτής, αλλά και ε, έλεγχο οποιασδήποτε διαδικασίας αποψήλωσης, ώστε κάθε μεμονωμένη ιδιοκτησία να διαφυλάσει κατά το 20% της ε, έκτασής της ε, την τροπική καλλιέργεια και επίσης να σέβεται τις, τις πηγές νερού. Και έτσι έχουμε καταφέρει να διαφυλάξουμε 80% της ε, του κάθε αγροτεμαχίου που βρίσκονται στην Αμαζονία. Ε, περιοχές που έχουν αποψηλωθεί στο απότερο παρελθόν εξακολουθούν να υποφελούνται από τη δυνατότητα διατήρηση το 50% των περιοχών ανάκτησης. Και η δική μας παραγωγικότητα απορρέει εν μέρη από τις, ε, από τις φυσικές συνθήκες, αλλά και από τις έρευνες και μελέτες που κάνουμε στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Έτσι καταφέραμε να έχουμε μια γεωργία που προσαρμόζεται στο τροπικό μας κλίμα. Πιστεύω ακράδαντα στις αρετές και τα πλεονεκτήματα του διεθνούς εμπορίου γιατί εκτός ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πιο ποιοτικά και πιο φθηνά προϊόντα στους καταναλωτές, θα μπορέσουν και οι χώρες να αξιοποιήσουν τους πόρους τους στις πιο παραγωγικές δραστηριότητες, αυξάνοντας τα εισοδήματα των γεωργών αλλά και την ε, κοινωνική ευημερία. Αλλά πέραν των αμυγός οικονομικών σχέσεων, το διεθνές εμπόριο φέρνει τους λαούς πιο κοντά και τους εντάσσει σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης ε, που είναι πολύ θετική και ανάρετη. Με ιδιαίτερη ε, ικανοποίηση. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την ισχυρή προσήλωση της Βραζιλίας στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων προκειμένου να δημιουργηθεί μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ του Μερκοσούρ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θεμελιώδης σημασίας για τη συνέχιση και διεκπαιρέωση των διαπραγματεύσεων να έχουμε ανταλλαγή προσφορών για την πρόσβαση στις αγορές αγαθών και ε, αυτές οι προσφορές να συγκεκριμενοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Στην αρχή της εβδομάδας ήμουν στην 83η συνέλευση του ΟΗΕ τη Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, Υγείας των Ζώων, όπου 12 πολιτείς της Βραζιλία, το Ρίο Γκράντζα του Σουλ και ε, οι δύο μάλλον της Βραζιλίας, Ρίο Γκράντζα του Σουλ και Σάντα Καταρίνα, αναγνωρίστηκαν διεθνώς ως ε, απαλλαγμένες από τον κλασικό ε, αυθόδη πυρετό το χείρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κτηνοτροφία μας και ευελπιστούμε ότι την επόμενη τριετία 14 επιπλέον πολιτείες της Βραζιλίας θα φτάσουν ε, σε αυτό σε αυτό το χαρακτηρισμό, δηλαδή θα τους αναγνωρίσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Ζώων ότι είναι απαλλαγμένες από τον αυτό πυρετό των πύρων. Το χείριο κρέας μας ε, που είναι ποιοτικό και διεθνώς αναγνωρισμένο Ελπίζουμε ότι θα φτάσει το συντομότερο δυνατό και στις ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης, ελπίζουμε ότι θα διεκπαιρεώσουμε τις ε, συμφωνίες με τις Ευρωπαϊκές Ακτινιατρικές Αρχές με βάση την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προσβλέπουμε σε μία ε, υγειονομική συμφωνία και ε, συμφωνία για κτηνιατρικά θέματα μεταξύ, και, μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διευκολυνθούν οι εμπορικές ροές ε, μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα διευκολύνουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές και τις εξαγωγές βοήου κρέατος και άλλων πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης η χώρα μου δεν είναι πλήρως ανοιχτή στο εμπόριο, το αναγνωρίζω. Και μεταξύ του πληθυσμού μας και των οικονομικών μας τελεστών, όπως και κάποιες χώρες άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, έχουμε και εμείς κάποια στοιχεία της νοοτροπίας μας που είναι δύσπιστα απέναντι στο εμπόριο. Ονειρεύονται μια οικονομική αυτονομία. Αλλά αυτά τα όνειρα είναι αυταπάτες, είναι σφαλμένα όνειρα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί το πεπρωμένο της σημερινής οικονομίας βρίσκεται στην υπέρβαση των εμποδίων και στην ολοκλήρωση. Η κατανάλωση ε, και η γεωργία έχουν γίνει οικομενικά φαινόμενα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, που μας ε, κρατούν όλους συνδεδεμένους. Επίσης, οι αλυσίδες παραγωγής δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα και διαρθρώνονται σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε προοδευτικοί, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει του ανοίγματο στον εμπόριο. Αυτή τη βδομάδα θα μεταβώ και στη Γενέβη και εκεί θα ε, διαμηνήσω το κατηγορηματικό μήνυμα ότι θέλουμε ενίσχυση του πολυμερού συστήματος του εμπορίου ε, που θα συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Θέλουμε πλήρη ενσωμάτωση της γεωργίας στο πολυμερέ σύστημα και επιθυμούμε ε, την ε, ολοκλήρωση του γύρου διαπραγματεύσεων της ΔΟΧΑΣ. Η, η Βραζιλιάνικη γεωργία δεν θα αρκεστεί σε μινιμαλιστικά αποτελέσματα στη διαπραγματεύση για τη γεωργία. Θέλουμε ε, επίσης ε, να δημιουργήσουμε και περιφερειακές εταιρικέ σχέσεις για να δώσουμε ένα νέο δυναμισμό στις οικονομίες και το εμπόριό μας. Ο παραγωγικός τομέας και η κυβέρνηση της Βραζιλίας αποδίδουν ύψιστη προτεραιότητα στην εμπορική συμφωνία της Βραζιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ώστε να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατόν στη σύναψη της συμφωνίας και ελπίζουμε ειλικρινά ότι τα θέματα της γεωργίας δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο στην διεκπαιρέωση αυτών των διαπραγματεύσεων. Ο γεωργικός προστατευτισμός, πολύ περισσότερο από τον βιομηχανικό, μπορεί να στερήσει ε, τον κόσμο ε, από σημαντικές παραγωγές ε, με απρόβλεπτες και αρνητικές συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα κατακλείδω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως είναι το καλύτερο πολιτικό οικοδόμημα του σύγχρονου ανθρώπου γιατί σε ένα αδελφικό πεπρωμένο συνένωσε λαούς που για αιώνες ολόκληρους ήταν ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Και αν κατέστη δυνατό αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, Σίγουρα πολλά πράγματα φαινομενικά αδύνατα ε, μπορούν κάποια στιγμή να, πραγμα... πραγματοποιηθούν. Αυτό πιστεύω και αυτή την αίσθηση έχω κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ μαζί με πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας ήταν ε, μεστή και αξιόλογη και τα λόγια σας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας άγγιξαν πραγματικά, μας συγκίνησαν. Χαιρόμαστε και εμείς και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζίλιας. Θα περάσουμε τώρα σε ένα γύρο των συντονιστών. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Άλμπερτ Ντες, που είναι ο συντονιστής ε, της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Υπουργό που ήρθε εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Γεωργίας. Χαίρομαι ιδιαίτερως. Ε, επί 10 χρόνια στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ήμουν ε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου με την Βραζιλία και έκτοτε με συνδέουν ε, σχέσεις φιλίας με πολλούς εκπροσώπους της ε, βραζιλιάνικης αντιπροσωπείας. Το Δεκέμβριο ήμουνα στο, στη Βραζιλία και το 88 είχα παραβρεθεί στη Βραζιλία. Πρέπει να σας συγχαρώ γιατί στη Βραζιλία έχουν αλλάξει πάρα πολύ προς τη θετική κατεύθυνση. Το 1988 διαπίστωσα ήδη πόσο μαζική ήταν η διάβρωση. Σήμερα λοιπόν ε, πρέπει να πω ότι πιστοποιώ ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες που, ε, που επικρατούν. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλη η κριτική που ασκείται στη Βραζιλία. 61% είναι δάση της έκτασης της Βραζιλίας και όποιος ε, περνάει με ε, αεροπλάνο το διαπιστώνει αυτό. Και δεν είναι μόνο οι παράνομες εταιρείε ηλεκτρομίας που δραστηριοποιούνται εκεί. 3.000 εκτάρια 700 εκτάρια τροπικού δάσους τα οποία είναι ανέπαφα αλλά και η υπόλοιπη επιφάνεια την οποία γνωρίζω εδώ και 26 χρόνια βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση παραγωγής. Αυτά που αναφέρατε, το εμπόριο, το διμερές, εδώ και οι δύο πλευρές θα πρέπει να επιτύξουν προθυμία. Κατά το παρελθόν έχω διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, το είπατε και εσείς άλλωστε, να εισάγουμε εμπορεύματα και προϊόντα προς την ε, Βραζιλία. Τεράστια είναι τα προσκόμματα σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, τα υλικά νοσοκομείου. Νομίζω ότι σε μία περίπτωση πήρε τέσσερις μήνες η εκτελεσμός τους. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτραπεί. Γι' αυτό λοιπόν και οι δύο πλευρές θα πρέπει να εργαστούμε για την άρση των εμποδίων. Αυτό που είναι το δικό μας πρόβλημα και είναι λιγότερο βρασιλιάνικο πρόβλημα είναι το εξή. Εμείς ε, επιβάλλουμε σαφή πρότυπα στους δικούς μας παραγωγούς. Αν τι γίνεται με τα πρότυπα αυτά στο υπόλοιπο του κόσμου. Δεν ήθελα να χρονοτριβήσω, αλλά θα ήθελα να επισημάνω αυτό που Έχω πει και στο παρελθόν και... Αν ήμουν 25 χρονών και ήμουν γεωργός, θα πήγαινα στη Βραζιλία. πλέον βέβαια είμαι πολύ ηλικιωμένος γι' αυτό. Σας εύχομαι καλή παραμονή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντές. Προσθέστε και μια προσωπική νότα στην ομιλία σας. Δεν ξέρω πώς επηγαίνατε, Με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο. Ο κύριος Δεκάστρο, πρώην πρόεδρος Επιτροπής Γεωργίας και πρώην Υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας. Ευχαριστώ πρόεδρε, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θέλω να σας καλωσορίσω κυρία Αμπρεού. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Το θέμα της ασφάλειας της προμήθειας τροφίμων στον κόσμο είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι μεγάλη πρόκληση να καλύψουμε τις ανάγκες ενός πληθυσμού που συνεχώς αυξάνεται στον τομέα των τροφίμων. Και αυτό περνά και από τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας σας τα τελευταία χρόνια. Η χώρα σας είναι η ηγέτης στις εξαγωγές πολλών γεωργικών προϊόντων, προϊόντων στα οποία εισάγει η Ευρώπη κυρίως όπως η σόγια. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και άλλη μια τεράστια προσπάθεια, το οποίο ξεκίνησε πειραματικά στη χώρα σας. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Φοντσίρο, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο μείωσε ε, την πείνα στην Βραζιλία. Και δεν ήταν μόνο θέμα κοινωνικής πολιτικής, αλλά επίσης ότι παράλληλα με τις κοινωνικές πολιτικές ακολουθήθηκαν και συγκεκριμένες πολιτικές στον τομέα της γεωργίας που επέτρεψαν αυτό το έκτακτο αποτέλεσμα το οποίο στην Expo 2015 στο Μιλάνο συζητάμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτό το σημαντικό σας επίτευγμα. Σας ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα γιατί τηρήσατε το χρόνο σας, γιατί ο κύριος Δες προηγουμένως τον υπερεύει. Ο κύριος Μουτσεχόφσκι τώρα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Νίκολσον. Ε, προς το παρόν ε, επιφυλάσσομαι. Δώστε σε άλλους το λόγο πρώτα. Η κυρία Μίλλερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για... Κλείνει δυστυχώς το μικρόφωνο της ομιλητρίας. Εγώ στην Βραζιλία ε, βρέθηκα το 2012 με αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κοινοβουλίου και εντυπωσιάστηκα από την εντατική καλλιέργεια της γης με βιώσιμο τρόπο και παράλληλα από την έκταση των καλλιεργειών και των βιοτόπων. Παρ' όλα αυτά, στη Γερμανία πάντα γίνεται η συζήτηση για την ε, η υλοτομία του τροπικού δάσους και σε ό,τι αφορά τα γενετικώ ε, τροποποιημένα προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται στη Βραζιλία. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω τρεις ερωτήσεις συγκεκριμένα. Εισαγάγουμε κυρίως ε, σπόρους γενετικώς τροποποιημένους. Ε, τι έκταση υπάρχει λοιπόν στην Βραζιλία με καλλιέργεια παραδοσιακών προϊόντων χωρίς γενετικά τροποποιημένα υλικά. Έχουμε μια βρία συνεργασία με την Βραζιλία, όπου μας αναφέρεται ότι η σόγια, η οποία δεν είναι γενετικώς ε, τροποποιημένη, εισαγάγεται. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Λέτε και μιλάτε για έρευνα και ανάπτυξη. Όταν μεταβήκαμε στη Βραζιλία, οι γεωργοί μας είπαν ότι σε ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση του κράτους για θέματα επιστημονικά καινοτομία, ουσιαστικά υποχρεούνται οι καλλιεργητέ να χρησιμοποιούν γενικώ τοποποιημένους σπόρους για να υπάρχουν μεγαλύτερη απόδοση. Ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να θίξω, τις διαπραγματεύσει με στα πλαίσια του TTIP μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν μειονεκτήματα για τους Βραζιλιάνους παραγωγούς και προωθείτε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Μερκουσούρ. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί είπατε ότι στην πατρίδα σας καταφέρατε να μειώσετε τη φτώχεια. Εδώ βρίσκομαι. Είμαι από τη Γαλλικία. Ε, και τα γαλλικιανά, ξέρετε, μοιάζουν πολύ με τα πορτογαλικά. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας ε, ενημερώσω ότι δυστυχώς ε, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης η φτώχεια αυξάνεται το ίδιο και η πείνα. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως να μου πείτε αν όντως το πρόγραμμά σας ε, ε, μηδενική πείνα, FOM 0, ανταποκρίθηκε στις προτεραιότητες και υλοποίησε τους στόχους σας. Επίσης, ε, τι γνώμη έχετε για το όνειρο των λαών να είναι αυτάρκες ό,τι αφορά τα βασικά προϊόντα διατροφής τους. Και το λέω αυτό κυρίως για τους λαούς της Αφρικής. Γιατί με αυτή την, αυτό το άγχος εξάπλωσης και ε, παραγωγής παγκόσμιας και από πλευράς Βραζιλίας αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στερούμε από πολλές χώρες τη δυνατότητα να παράγουν τα δικά τους τρόφιμα. Είπατε ότι στόχος σας είναι να εξαγάγεται χείριο και βόλιο κρέας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για τη σοβαρότατη κρίση που ε, βιώνουν αυτή τη στιγμή η γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κτηνοτρόφη εξαιτίας ε, του ρωσικού εμπάργου στις εισαγωγές προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς τις μικρομεσαίες γεωργικές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις απέναντι σε αυτές τις τρομερές διακυμάνσεις που προκαλούν οι εξαγωγές. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και εγώ. Είχα πάει πέρυσι στην ωραία σας χώρα και μου έκανε εντύπωση ο πλούτος των φυσικών πόρων και τα μέτρα, ε, τα, μέτρα τα οικολογικά και ε, μέτρα που στοχεύουν στην αηφορία γενικότερα τα οποία έχετε πάρει. Είχα πάει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα συζητηθούν και στη συνάντηση κορυφής για το κλίμα στο Παρίσι. Η Βραζιλία όπως όλες οι χώρες υποφέρει τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης υδάτινων πόρων. Η 34η έκθεση της Λέσχης του Ρώμου, λέγει, της Ρώμης, συγγνώμη, λέγει ότι ε, στον τομέα των υδάτων, στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα της γεωργίας τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον. Εγώ προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη χώρα που οδήγησε τον κόσμο ε, στην βιομηχανική επανάσταση και νιώθω μια κάποια ευθύνη για τις εκπομπές καυσαερίων και για την ανάγκη που υπάρχει για τη Βραζιλία να προστατεύσει ε, τα τροπικά δάση και επίσης και τις δασικές περιοχές γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Σαν πλούσια πλέον και ισχυρή χώρα θα παίξετε ένα σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι. Η αδίποτε συμφωνία θα είναι στην ουσία ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στις μεγάλες χώρες και τις χειρές οικονομίες που κληρονόμησαν καθαρά περιβάλλοντα τα οποία φυσικά ε, βοηθούν την αντιμετώπιση των συνεπειών της εκπομπής καυσαίριων. Η κυβέρνησή σας έχει προτάσεις συγκεκριμένες και τι περιμένει έτσι ώστε να πάρει μέτρα για να διασωθούν ε, περισσότερα τμήματα της ε, δασικής περιοχής του Αμαζονίου. Σας ευχαριστώ κύριε Άγνιου. Well, good afternoon, Minister. Καλησπέρα Υπουργέ και θα σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι η αναφορά της χώρας σας, Βραζιλίας, ε, προκαλεί φόβους, μπορεί και τρομοκρατία, τρόμο στην ε, χώρα μου. γιατί πρόκειται για μια χώρα με πάρα πολλές εκτάσεις όπου ε, υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν είναι υψηλότερο το εργατικό κόστος και μπορεί κανείς να παράγει μέχρι και δύο σοδιές κάθε χρόνο. Ήδη εξαρτώμαστε από εσάς για την πρωτεΐνη μας, από τη σόγια και θα θέλαμε να μας πείτε από πολιτικής άποψης τι ισχύει και πώς μπορείτε να αποκριθείτε στις ανησυχίες μας. Αναφερθήκατε στον θέμα της γρήπης των χείρων ανάλυση των χείρων και των μαζικών τέτοιων ε, επιζωτιών. Ε. Αυτό δυσπηρετός από ό,τι καταλαβαίνετε εξακολουθούν να υπάρχουν και να πλήττουν τη Βραζιλία. Έχουμε τεράστια προβλήματα στη χώρα μου πριν από 14 χρόνια και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κανένα του περιορισμού. Τέλος, δεν πιστεύω ότι η χώρα σας έχει σταματήσει τη χρήση κλωβών για την παραγωγή αυγών. Μάλλον θα έλεγα ότι εξαρτάστε από αυτά. Όπως ξέρετε, αυτό δεν επιτρέπεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι λοιπόν η στάση σας και τη μετώπιση σας. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο ε, τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Βραζιλία, τον κύριο Ζωρίνιο. Ευχαριστώ. Ως Αντιπρόεδρος της ε, Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Βραζιλία θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ. Οι σχέσεις ε, Ευρώπης-Βραζιλίας και ιδιαίτερα οι σχέσεις Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής έχουν τεράστια στρατηγική σημασία. Επίσης, ε, ε, η επίσκεψή σας πραγματοποιείται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη Eurolat, τη Συνέλευση Ευρώπης Λατινικής Αμερικής και τη μέθε επόμενη εβδομάδα θα έχουμε στη Βρυξέλλες τη διακυβερνητική ε, διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΑΚ. Οπότε επίκαιρη η επίσκεψή σας για να ξαναθέσουμε σε νέα ισορροπία το, τα διάφορα στοιχεία η διαδικασία της παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε από τους Άγγλους με τη βιομηχανική επανάσταση όπως είπε η συνάδελφος. Θα πρέπει να δούμε όμως και τις πολιτικές αξίες, ανθρωπιστικές αξίες, πολιτιστικές αξίες που είναι κοινέ μας αξίες και χαρακτηριστικά της κοινή μα ταυτότητας. Η Ευρώπη και η Βραζιλία έχουν συγκλίνοντα στρατηγικά συμφέροντα παρά τις διαφορές τους. Θα πρέπει να αυξήσουμε, είπατε, τις εμπορικές συναλλαγές, να διαφοροποιήσουμε τις αγορές μας, να ελαφρύνουμε τους ε, φραγμούς, να επενδύσουμε στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και στην εφόρο ε, ανάπτυξη. Έχουμε τις πιο ανεπτυγμένες ε, γεωργικές δομές του κόσμου και τα προϊόντα μας είναι δυνάμει προϊόντα εξαγωγής. Υπάρχουν όμως και κάποιες ζώνες ανταγωνισμού μεταξύ μας και κάποια επίμαχα σημεία σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές και τα πρότυπά μας. Θα συμφωνείτε όμως μαζί μου ότι η λύση για να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας και όλα αυτά τα θέματα ε, και να άρουμε τους φραγμούς στη συνεργασία θα πρέπει να καταλήξουμε σε συνολική σφαιρική λύση. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να διεκπαιρεώσουμε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση και Μερκοσούρ. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσα την προσήλωση και τη δέσμευσή σα για την αίσια διεκπαιρέωση αυτή τη συμφωνία. Βέβαια, ε, υπάρχουν πολιτικές δυσκολίε ε, ε, σε κάποιες χώρες του Μερκοσούρ και το ίδιο και στις κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική και δύσκολη αυτή η πρόκληση. Θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν αποφασιστικότητα και πολιτικό θάρρο για να φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτή τη συμφωνία και ελπίζω η επίσκεψη να στεφθεί με επιτυχία και για τι δύο περιοχέ μα και να διεκπαιρεωθούν αισίω οι διαπραγματεύσει με τη Μερκοσούρ. Ευχαριστώ και βάζω τελεία εδώ κύριε Πρόεδρε. Dalsze wypowiedzi pani Σας θέρμα παρακαλώ υπόλοιπα να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Ρεμπέγκα. Oh, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλώς ορίσατε την κυρία Υπουργό. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις να θέσω. Δεδομένου του ότι η Βραζιλία αποτελεί έναν από το βασικό παραγωγό γενετικώς τροποποιημένων ε, φυτών, σόγιας και δεδομένου επίσης ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένου λοιπόν ότι η Βραζιλία παράγει σε μεγάλη κλίματα, κλίμακα σόγια, γενετικώς τροποποιημένη. Και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισαγάγει τη σόγια αυτή. πώς θα σας φαινόταν να εναρμονιστείτε με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι φέτος θα πρέπει να αποφασίσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πόσον ε, θα επιτρέψουν ή όχι την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένης ε, σόγιας. Κάτι άλλο. Για να υποστηρίξουμε τους νεαρούς ε, αγρότες. Θα το σκεφτόσασταν αυτό. Στη Βραζιλία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σα ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συνάντηση αυτή. Σας ευχαριστώ επίσης και για τις πολύτιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Ε, κάποιες ερωτήσεις θα ήθελα. Καταρχάς, οι συνέπειες της μεταρρύθμισης της αγοράς της Ζάκαρης. Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε αυτές τις αλλαγές για να περιορίσουμε την παραγωγή ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είχε τεράστιες συνέπειες στους Ευρωπαίους γεωργούς. Θα ήθελα να μάθω αν έχουν υπάρξει επιπτώσεις στην αγορά και στην παραγωγή του προϊόντος αυτού στην Βραζιλία. Υπήρξε αύξηση των αμοιβών των γεωργών, αυξήθηκε η παραγωγή, ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι ζαχαροπαραγωγές. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη, το θέμα της ε, ευημερίας των ζώων, το θέμα της ευζωίας. Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Το λαμβάνετε υπόψη στην κτηνοτροφία σας, στο θέμα της ευζοίας. Και έχετε προδιαγραφές για τα θέματα της ευημερίας των ζώων. Τραβάει καθόλου την προσοχή της κυβέρνησης Βραζιλίας σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριο Σμιθ. Uh, uh, σας ευχαριστώ. Και εγώ έχω πάει στη χώρα σας ε, πέρυσι πήγαμε στις εκτινοτροφικές περιοχές, στο Ματογκρόσο και στο Νότα, είδαμε τι συμβαίνει εκεί, συγκρίναμε με αυτά τα οποία γίνονται στη Σκοτία και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τα υψηλά επίπεδα κατάρτισης των γεωργών σε τομέα όπως η γενετική κτλ. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Βέβαια οι εμπορικές συναλλαγές θα πρέπει να βασίζονται σε δίκαια και ισότιμα επίπεδα. Θα ήθελα εδώ να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Άγνιου για τις, ε, ε, για διαδικασίες εμβολιασμού στην περίπτωση του Αθόδους. Και επίσης θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται με την κυριαρχία την οποία πρέπει να έχει μια περιοχή και μια χώρα στον τομέα των τροφίμων ε, δεν μπορεί εμείς να επαφιέμεθα σε άλλες αγορές για τις προμήθειες. Ε, εσείς στην ε, Βραζιλία με συγκεκριμένες δανειοδοτήσεις και συγκεκριμένες δραστηριότητες διασφαλίσατε την επάρκειά σας στην διατροφική. Μήπως πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ. Ε, η Βραζιλία είναι μια μεγάλη χώρα που νόμιμα θέλει να καταλάβει άλλες αγορές αλλά σαν ε, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας της Γαλλίας είμαι κατά των προϊόντων γενετικά τροποποιημένων. Ε, εμείς απορροφούμε το 58% της σόγιας για τις κτηνοτροφές ιδιαίτερα στον βόρειο τομέα και επίσης και στον τομέα της παραγωγής χείριου κρέατος κατά 12%. Ε, οι επιφάνειες παραγωγής ε, σόγιας έχουν 20 ε, πλασιαστεί σε 40 χρόνια. Είστε ο έκτος παραγωγός επίσης διοξιδίου του άνθρακος. Η πολιτική σας συνοδεύεται από την παρουσία πολιεθνικών στην χώρα σας θυγατρικών από τις Ηνωμένε Πολιτείες, ιδιαίτερα που ασχολούνται με τα γενετικά χαρακτηριστικά της, των πτηνών. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις προς την κυρία Μπρέου. Τι ισχύει στην Βραζιλία στον τομέα της χρήσης των αυξητικών ορμονών για το βόηο κρέας και ποιο είναι το κόστος δεύτερον της παραγωγής βοήου κρέατος γενικότερα. Κύριε Νταντσίλα. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια και για αυτή την λεπτόμερη και παθιασμένη παρουσίαση. Δεν έχω επισκεφτεί τη Βραζιλία, αλλά θεωρώ ότι η ανταλλαγή των πρακτικών αποτελεί α, κάτι το απαραίτητο, γιατί είσαστε και παγκόσμιο ηγέτη τη ε, εξαγωγή. έχω διαπιστώσει ότι οι γυναίκες στη χώρα σας με τον υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και επαγγελματισμού συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχουν ε, σταθεροποιητικό ρόλο και προωθούν τον εξυγχρονισμό στον κλάδο αυτό. Πώς ε, θεωρείτε λοιπόν ότι διαμορφώνεται ο ρόλος της γυναίκας στην ε, γεωργία και τι θα πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, τι αξιώσεις πρέπει να θέσουν για να διασφαλίσουν τον ρόλο τους. Προβλέπετε κάτι στο πρόγραμμα σας περαιτέρω. Ο κύριος ε, Καλώς ορίσατε εδώ στο Κοινοβουλίο, κυρία Υπουργέ. Μας δείξατε ότι η παραγωγικότητα στην Βραζιλία έχει αυξηθεί, αλλά δεν πιστεύετε ότι το θέμα της διανομής είναι το πρόβλημα βασικά. Και όχι μόνο η αποκλειστική αύξηση της παραγωγής. Ένα δεύτερο θέμα που αφορά την κατανομή. Η ανισόρροπη κατανομή της γης είναι ένα πρόβλημα στη χώρα σας και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Και η καλλιέργεια ημί της ε, γης θα ήσασταν ε, διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη χρήση της γης προκειμένου να λάβουν ιδιαίτερη υποστήριξη και οι μικροκαλλιεργητές γιατί αυτοί συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον επισητισμό της γης μας. Αναφερθήκατε στο μεγάλο τμήμα της έκτασης που διατηρούν την φυσική τους κατάσταση αλλά πιστεύετε ότι είναι επαρκής αυτή η διατήρηση του Αμαζονίου ή χρειάζονται και περαιτέρω μέτρα. Μία ερώτηση επίσης θα ήθελα να θέσω περαιτέρω. Πιστεύετε ότι στο μέλλον οι Ευρωπαίοι στο μέλλον θα συνεχίσουν να εισαγάγουν γενετικώς τροποποιημένη σόγια και πιστεύετε ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική υποστήριξη του μελλοντικού μας εμπορίου. Ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 ε, θέσπισε ως ε, στόχο ε, την αύξηση κατά 10% των βιο... της βιομάζας και της μεθανόλης με τα βιοκαύσιμα θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να εξασφαλίσουμε γεωρικά εισοδήματα. Πριν από τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε ε, αναθεώρηση της χρήσης ε, των γεών και μείωσε κατά το ίμιση το στόχο. Η, η Βραζιλία είναι, από τις... είναι ο πρώτος εξαγωγός παγκοσμίως βιοκαύσιμα και κυρίως μεθανόλης. Ε, βέβαια, μερικές φορές αυτό γίνεται εις βάρος σημαντικών βιοτόπων ε, για το περιβάλλον. Πώς βλέπετε αυτό, αυτή την αλλαγή της χρήσης γης ε, προκειμένου να παραχθούν και να διονυστεί η παραγωγή βιοκαυσίμων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Υπουργέ που μας παρουσιάζετε τη γεωργία της χώρας σας και προασπίζεστε τη γεωργία της χώρας σας. Αναφερθήκατε επίσης στις διεθνείς συναλλαγές. Η Βραζιλία πιστεύει άραγε ακόμα στον ΠΟΕ. Η ίδια η Βραζιλία έχει ξεκινήσει με τις διμερείς συμφωνίες. Θεωρείται ότι ο γύρος της Ντόχα υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί στον τομέα της γεωργίας ποτέ. Ο κύριος Yeah. κυρία μου. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Στην Ευρώπη έχουμε το εκτή πρόβλημα. Οι επιδοτήσει ε, κυρίως χορηγούνται στι μεγάλε επιχειρήσει αλλά στη Βραζιλία ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την έκθεση του ΑΣΕ για τις άμεσες επιδοτήσεις. Η πληρωμή 2004 από 3 δισεκατομμύρια το 2010 έφτασε τα 10 δισεκατομμύρια και αυτό ασφαλώς υποτελεί ε, αντικείμενο κερδοσκοπίας. Είσαστε μεγάλο κτηματίας ουσιαστικά στη Βραζιλία. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρυθμίσης και τη συμπερίληψη τη συνεργασία σε θέματα απασχόληση στην Ήπεθρο. Έχατε έναν υπουργό στην ε, Βραζιλία για την ανάπτυξη της Υπέτρου. Υπάρχει γενικώ ομοφωνία και συνένεση για αυτά που επικρατούν στη Βραζιλία ή μήπω ε, εξετάζεται το ενδεχόμενο ακολούθηση ενό διαφορετικού δρόμου. Pan, pan Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Υπουργέ για το γεγονός ότι ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω μετά τους συναδέλφους για τη γενετικώς τροποποιημένη τεχνολογία. Τι γίνεται με την κοινωνική, τον κοινωνικό διάλογο για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους. Πώς είναι η κατάσταση στη χώρα σας, πώς συζητιέται το θέμα ένα άλλο θέμα για την χρήση των φυτικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας, εθανόλης. Πώς διεξαγάγει τη συζήτηση. Και τρίτη ερώτηση. Και εδώ στην Ευρώπη γίνεται η συζήτηση για τους μικρούς ή μεγάλους καλλιεργητές. Υπάρχει τέτοια, τέτοιος ορισμός στη χώρα σας. Τι θεωρείτε σε εσάς μεγάλος ε, καλλιεργητής και τι θεωρείτε μικρός. Ο κύριος Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον ε, όλα αυτά που άκουσα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν έχω μεταβεί ποτέ στη χώρα σας, αλλά επειδή μου απασχολεί και το θέμα του αποτυπώματος του άνθρακα, μάλλον δεν πρόκειται να επισκεφτώ και τη χώρα σας ποτέ. Εγώ στη δική μου χώρα ακούω και από άλλες χώρες ότι θέλουμε να δώσουμε τρόφιμα σε όλο τον κόσμο. Είναι ασφαλώς πάρα πολύ ε, θεμητό και φιλόδοξο αυτό στόχος, αλλά κάποιες χώρες απλά θέλουν να πλουτίσουν. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς γι' αυτό. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο αν μπορούσαν οι χώρες να θρέψουν τον ίδιο τους το πληθυσμό. Και επίσης, αν ε, καταφέρετε να εξαγάγετε πιο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς αυτό θα βλάψει τους δικούς μας καλλιεργητές και παραγωγούς. Πώς λοιπόν, ρωτιέμαι, πρόκειται αυτό να μας ωφελήσει. Και τέλος, ήταν εξαιρετικές οι ερωτήσεις που ετέθησαν και ανυπομονώ να ακούσω τις απαντήσεις, αλλά είπατε πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το πιο όμορφο πολιτικό οικοδόμημα που υπάρχει, γιατί εγώ σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ με αυτό. Każdy słyszy, co chce słyszeć ο καθένας ακούει αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν βλέπω άλλο να ευρωβουλευτή να ζητά το λόγο. Α, συγγνώμη, κύριο Σεμπαστιά. Ο κύριος Σεμπαστιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Η ερώτηση δεν είναι δικιά μου. Ε, από κάποιους ε, φίλους από το Μάτο Γκρόσο ε, μου στείλαν την ερώτηση. Ε, να μιλήσουμε για την ιδιοκτησία των γεών. Πάνω από 25 χρόνια γνωρίζω αυτούς τους φίλους μου που είναι ηθαγενείς, ε, ακτήμονες και μάλιστα έχασαν ε, τη, τα εδάφη τους εξαιτίας των φαζεντέρων, των μεγάλων ε, γεωκτημόνων. Και 25 χρόνια μετά δεν έχουν ανακτήσει αυτές, ε, αυτά τα χωράφια που είχαν. Τι θα κάνει το Υπουργείο σας για να επιστρέψουν τα χωράφια στους ακτήμονες, ε, σε αυτούς που παραδοσιακά καλλιεργούν αυτά τα εδάφη, για να επανέλθουν και να ανακτήσουν τα δικαιώματα τους ηθαγενείς και όλοι αυτοί οι γεωργοί που έχασαν τα, τα χωράφια τους. Ευχαριστώ. Ε, Και ο κύριος Μποβέ είναι ο τελευταίο μας ομιλητής. Υπουργέ καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Έχω πάει επανειλημμένα στη Βραζιλία. Έτσι μπόρεσα να πάρω μέρος σε πολλές δραστηριότητες όπως την καταστροφή των γενετικά τροποποιημένων λιβαδιών της Μονσάντο μαζί με το κίνημα των αστέγων, των ακτιμώνων μάλλον. Θέλω δύο θέματα να θέσω. Πρώτον, φοβάμαι ότι μετά από αυτά τα οποία ακούμε, η Βραζιλία στην ουσία είναι το αεροπλανοφόρο της βιομηχανίας κρέατος, ιδιαίτερα στο χοιρινό κρέας και στα κοτόπουλα. Για πάρα πολλά χρόνια η Ευρώπη εκμεταλλεύτηκε τη Βραζιλία, ιδιαίτερα την εταιρεία Ντούγκ, η οποία είχε μεγάλη παραγωγή στη χώρα σας, ευτυχώς σταμάτησε. Θα πρέπει όμως οι αγορές να ανταποκρίνονται κυρίως στις τοπικές διαστάσεις και όχι σε λογικές εκμετάλλευσεις. Μια δεύτερη ερώτηση, πιο συγκεκριμένη για ένα δράμα σημαντικό στη Βραζιλία. Πέρα από το θέμα της γης, για το ρόλο της ευκαλύπτου. Η ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο της ε, φυτείας από ευκαλύπτους ε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα διότι διώχνει τους γεωργούς και αποστηρώνει τις γέες. Νομίζω ότι τώρα πια έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των ομιλητών. Και τώρα θα μπορούσαμε να ξαναδώσουμε το λόγο στην Υπουργό. Δεν ξέρω τι είναι ευκολότερο για σας. Ήταν, είναι πιο εύκολο να απαντάτε ερωτήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη οι συμπατριώτες σας στην εθνική σας βουλή, στη Βουλή της Βραζίλιας. Πάντως όλα υποβλήθηκαν με φιλικό πνεύμα και σε φιλικό κλίμα. Εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων, όπως καταλάβατε. Ακούσατε τις ερωτήσεις, ακούσατε τα σχόλια. Έχετε τώρα την ευκαιρία να απαντήσετε όπως επιθυμείτε και όσο επιθυμείτε. θα χρειαζόμαστε πραγματικά πάρα πολύ χρόνο για να απαντήσουμε σε όλες ε, τις ερωτήσεις. Ε, χρόνο που αξίζει να αφιερώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί οι ερωτήσεις ήταν πολύ σημαντικές και θα ήθελα να έχω πολύ περισσότερο χρόνο για να απαντήσω διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις ε, και θα το έκανα με ιδιαίτερη χαρά μάλιστα. Θα προσπαθήσω, χωρίς να ακολουθήσω τη συγκεκριμένη σειρά της υποβολής των ερωτήσεων, να επικεντρωθώ σε ορισμένες από αυτές. Καταρχήν, για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, τα μεταλλαγμένα και ιδιαίτερα τη μεταλλαγμένη σόγια. Ε, Οχτώ χρόνια ήμουν γερουσιάστρια, τέσσερα χρόνια βουλευτή, δώδεκα χρόνια δηλαδή συνολικά και πριν από 15 χρόνια είχαμε τεράστια δυσκολία στη Βραζιλία για να εγκρίνουμε τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Ήταν ε, δύσκολο να δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει ε, τι γίνεται με τα προϊόντα αυτά. Και εμείς οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί είμαστε απόλυτα έτοιμοι και πρόθυμοι να καλύψουμε τις ανάγκες αγοράς. Δεν έχουμε ε, παραγωγούς που ε, παράγουν γενετικό τροποποιημένους οργανισμούς για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θέμα της τιμής των ε, τροφίμων. Φυσικά η υγεία του ανθρώπου βρίσκεται στη βασική, ως βασική προτεραιότητα, αλλά και η υγεία των τροφίμων, η ασφάλεια των τροφίμων. Γιατί όταν μιλούμε για τον περιορισμό των καλλιεργήσιμων ε, γεών σε όλες τις περιοχές του κόσμου, για μας, ε, για την πλειοψηφία τουλάχιστον των Βραζιλιάνων, οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί είναι λύση, δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι ε, εμπόδιο τα μεταλλαγμένα για μας, αλλά μία ευκαιρία για αύξηση της παραγωγής με χρήση λιγότερων φυτοφαρμάκων γιατί αν, εφαρμοστούν καταχρηστικά και τα φυτοφάρμακα μπορούν να πλήξουν την ανθρώπινη υγεία και να είναι επιζήμια. Επίσης, με την ε, χρήση των φυτοφαρμάκων αυξάνεται και το κόστος παραγωγής. Για παράδειγμα, το μαβάκι που καλλιεργούμε ε, στην ε, Βραζιλία. Θα θυμάστε ότι εμείς ε, διαβιών, ε, ζούμε και παράγουμε σε μια τροπική χώρα. Δεν είμαστε σε, ευρωπαϊκό κλίμα. Εμείς έχουμε ζυζάνια και ε, φυτικές νόσους που θα πρέπει να αντιμετωπιστούμε ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα. Στο βαμβάκι, για παράδειγμα, αν καλλιεργούσαμε, αν φυτέβαμε το παραδοσιακό βαμβάκι, την παραδοσιακή ποικιλία βαμβακιού, θα είχαμε αύξηση του κόστους παραγωγής ε, που θα έβγαζε τη Βραζιλία πλήρως εκτός παγκόσμιου ανταγωνισμού. Θα έπρεπε να ε, σταματήσουμε την παραγωγή βραζιλιάνικου βαμβακιού. Εμείς, χάρη στα μεταλλαγμένα, μειώσαμε περίπου κατά 50% τη χρήση φυτοφαρμάκων στην παραγωγή βαμβάκιου. Οπότε χάρη στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς καταφέραμε να μειώσουμε τους ψεκασμούς με φυτοφάρμακα. Βέβαια, εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις και καταλαβαίνω και αυτούς που φοβούνται τα μεταλλαγμένα, άλλους όμως που είναι υπέρ των μεταλλαγμένων, αλλά μην ξεχνάτε και τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν σαφή αποτελέσματα. Και αν αναλύσουμε την παγκόσμια κοινωνία τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε ότι κάθε χρόνο, την τελευταία 20 ετία, έχουμε κερδίσει τρεις μήνες ζωής επιπλέον σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής. Οπότε σε ολόκληρο τον κόσμο παρόλο που ε, χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα, παρόλο που χρησιμοποιούμε μεταλλαγμένα, παρόλα αυτά δεν μειώνεται το προσδόκιμα της ζωής, αλλά αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Αυτό δεν είναι σημαντικός δείκτης. Οι παππούδες μου ε, και οι πιο ειλικρινοί λένε ότι η υγεία περνάει από το στόμα. Ό,τι τρώμε ε, καθορίζει την υγεία μας. Οπότε αυτή την άποψη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα εργαζόμαστε με βάση τις ανάγκες αγοράς. Εφόσον η αγορά αποδέχεται τα μεταλλαγμένα, εμείς τα προτιμούμε. Γιατί το κόστος της παραγωγής μας μειώνεται χάρη στα μεταλλαγμένα. Τώρα, αν μία χώρα θέλει να καταναλώνει ε, μη μεταλλαγμένα προϊόντα ή χωρίς φυτοφάρμακα, γιατί δεν είναι συμβατά μεταξύ τους, θα πρέπει να λάβει υπόψη το κόστος που συμπεριλαμβάνεται στην παραγωγή. Όσοι ε, δίνονται και θέλουν να πληρώσουν αυτή τη διαφορά και να πληρώνουν πιο ακριβά τα τρόφιμά τους, έχουν απόλυτο δικαίωμα να το κάνουν. Αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν έχουν όλοι την πολυτέλεια να ε, λαμβάνουν υπόψη τις προκαταλήψεις τους μερικές φορές. Γι' αυτό και θα πρέπει να ακούσουμε την επιστήμη. Οι επιστήμονες θα πρέπει να μας πούν τι επιτρέπεται και τι όχι. Εμείς γνωρίζουμε τα απορίσματα των επιστημόνων. Οι η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων σχεδόν σε όλες τις υπήρους δεν βλέπουμε κακό μάτι τα μεταλλαγμένα. Γι' αυτό και αυξάνεται η κατανάλωση και των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και ταυτόχρονα του προσδόκιμου ζωής σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας πω ότι και επανέρχομαι εδώ σε μεμονωμένα θέματα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πίνα 0, φόμη 0, πολλοί ρώτησαν πώς κατάφερε η Βραζιλία να φτάσει εδώ που έφτασε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν κάναμε μαγικά. Η Βραζιλία, χάρη στη φορολογική της ισορροπία και στην εφαρμογή ενός ρεαλιστικού σχεδίου, κατάφερε να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό και οι προηγούμενε κυβερνήσεις του Φερνάντε και μετά του Πρόεδρου Λούλα και τώρα με την Ντίλμα Ρουσέφ όλες οι κυβερνήσεις έμειναν στη φορολογική προσαρμογή, στην δημοσιονομική εξυγίαση, προκειμένου να ελέγξουν τον πληθωρισμό. Ακριβώς επειδή εφαρμόσαμε τον έλεγχο του πληθωρισμού και την δημοσιονομική προσαρμογή καταφέραμε στην Βραζιλία να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και μάλιστα το πρόγραμμα αυτό δεν το λέμε πια πίνα μηδέν, αλλά ε, το ε, ε, λέμε ένα επίδομα για την οικογένεια. Είναι ένα συμπλήρωμα ώστε οι άνεργοι ή όσοι βγάζουν λιγότερο από 70 ρεάις σαν μέλος της οικογένειας να μπορούν να λαμβάνουν αυτό το συμπληρωματικό επίδομα. Αυτές, αυτές ήταν οι επιλογές τριών διαδοχικών κυβερνήσεων που κάθε μία κράτησε, είχε θητεία οκταετή. Μιλούμε για δεκαετίες ε, εφαρμογής της ίδιας πολιτικής καταπολέμησης του πληθωρισμού και συμπληρώματος του εισοδήματος προκειμένου να φτάσει η μικρο μεγαλωστική τάξη στη μεσαία. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού μας στη μεσαία τάξη σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα. Και το, η νέα μας πρόκληση είναι και στις αγροτικές ζώνες και ε, στην Ήπεθρο που έχουμε 12 εκατομμύρια κατοίκους και 5 εκατομμύρια παραγωγούς να μην έχουμε την ίδια κατάσταση και μάλιστα μαζί με τις οικογένειες θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε 20 εκατομμύρια στην Ήπεθρο. Έχουμε ακόμη ε, τάξεις Δ και Ε αρκετά μεγάλες και τάξεις Α και Β σχετικά μικρές. Και έχουμε και μια μεσαία τάξη που οφείλει να διευρυνθεί, να μεγαλώσει. Τώρα ξεκινάμε ένα σημαντικό πρόγραμμα στη Βραζιλιάνικη κυβέρνηση για να διευρύνουμε αυτή την Βραζιλιάνικη μεσαία τάξη για να έχει και αυτή η μεσαία τάξη πρόσβαση στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην τεχνική αρρωγή και στην, στην επαγγελματική κατάρτιση. Για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς επίσης να ε, οργανώνονται. Γιατί ο καθένας μόνος του και ε, με δυσμενείς όρους θα αγοράζει και με δυσμενείς όρους θα πουλά. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να οργανώνονται σε συνεταιρισμούς η παραγωγή, ώστε να μπορούν να αγοράζουν τις πρώτες ύλες τους μαζί και ταυτόχρονα να διαθέτουν τα προϊόντα τους από κοινού σε ευνοϊκότερους όρους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία της γης. Η μέση ιδιοκτησία ε, επαναλαμβάνω, έχουμε 5 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Από αυτές ε, η μέσος όρος είναι 67 εκτάρια. Ε, η Βραζιλία με 85 εκατομμύρια εκτάρια έχει 5 εκατομμύρια παραγωγούς. 5 εκατομμύρια παραγωγούς. Αν προσθέσουμε και τον Καναδά και τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Αυστραλία μαζί, δεν φτάνουμε ούτε σε 3 εκατομμύρια. Έχουν 2.700.000 ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ στη Βραζιλία έχουμε 5 εκατομμύρια. Οπότε έχουμε μια πολύ ορθολογική κατανομή των ε, γεών και των εδαφών στη Βραζιλία. Για παράδειγμα, 10% όλης της παραγωγικής έκτασης της Βραζιλίας βρίσκεται στα χέρια γεωκτημόνων από τη γεωργική μεταρρύθμιση, ένα πολύ παλιό πρόγραμμα κατανομής των γεών στη Βραζιλία. 10% δηλαδή 80 εκατομμύρια εκτάρια βρίσκονται στα χέρια μικρών καλλιεργητών με βάση αυτό το πρόγραμμα και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Η παραγωγή αυτή δικαίως έλαβαν ε, τα χωράφια αυτά από την κυβέρνηση. Δυστυχώς η κατάσταση της συντριπτικής πλειοψηφία αυτών των καλλιεργητών δεν είναι πολύ ευνοϊκή. Θα πρέπει να βελτιωθεί το γεωργικό του εισόδημα γιατί η κατάστασή τους προς το παρόν είναι δεινή ώστε να μπορέσει πραγματικά η γη να τους ε, ωφελήσει και να συμβάλλει στην αύξηση του γεωργικού του εισοδήματος. Γιατί ουσιαστικά η πρώτη σύλληση για τη γη είναι 15 με 20% τη γεωργικής παραγωγής. Το υπόλοιπο είναι έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, εργατικό δυναμικό, ε, επαγγελματικά προσόντα. Αλλά το αγροτεμάχιο, το χωράφι το ίδιο, και αυτό το λέω στα παιδιά μου που θα με διαδεχτούν στο αγρόκτημα, η γη, το αγροτεμάχιο είναι απλώς η αρχή του προβλήματος. Έχουμε και πολλά άλλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Πάντως πιστεύουμε ότι 80 εκατομμύρια εκταρίων που διανέμονται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, σε, μικρά, σε μικρές καλλιέργειες και από αυτό το τεράστιο πλαίσιο γεωργίας και κτηνοτροφίας, ε, εμείς μόνο σε 50 εκατομμύρια εκτάρια φυτεύουμε ε, και χρησιμοποιούμε για την εκτροφή των ζώων. Και επαναλαμβάνω, 10% του, της επικράτειας είναι από το πρόγραμμα της γεωργικής μεταρρύθμισης και 6% αυτών των 5 εκατομμυρίων παραγωγών είναι μικροκαλλιεργητές με τέσσερα ε, με τέσσερις μόνο φορολογικές μονάδες ουσιαστικά γη, δηλαδή περίπου 320 εκτάρια ε, ανήκουν στον κάθε μικροπαραγωγό, που είναι 86% επαναλαμβάνω του συνόλου των βραζιλιάνων παραγωγών, που είναι συνολικά 5 εκατομμύρια. Από τα 5 αυτά εκατομμύρια, το 86% είναι μικροκαλλιεργητές. 12% είναι η μεσαίη παραγωγή από αυτά τα 5 εκατομμύρια. Αυτή η μεσαίη παραγωγή έχουν 4 με 15 φορολογικές μονάδες, δηλαδή 1200 εκτάρια το πολύ, αυτή η μεσαία παραγωγή. Τέλος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε στον κόσμο ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα λατιφουντίων και φέουδων. Έχουμε μεγάλες καλλιέργειες, αλλά δεν είναι, δεν είναι αντιπαραγωγικές. Σίγουρα κάποιες ζώνες θα πρέπει να βελτιώσουν την παραγωγή τους και έχουμε και περιοχές όπου ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τα εισοδήματά τους, αλλά δεν υπάρχουν αντιπαραγωγικές εκτάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιβίωση των χωρών και την αυτάρκεια σε τρόφιμα από την παραγωγή, εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό όλες οι χώρες που θα πρέπει να έχουν τη δική τους παραγωγή. Και όσοι ε, μπορούν να το κάνουν, μακάρι να το πετύχουν και χειροκροτώ και επικροτώ αυτό το όραμα. Πριν μάλιστα από 40 χρόνια, τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 60 λοιπόν, η Βραζιλία ε, ήταν αναγκασμένη να εισάγει το, με, μεγαλύτερο τμήμα των τροφίμων ε, ε, ρύζι από τις Φιλιππίνες, ε, γάλα από την Ευρώπη, φασόλια από το Μεξικό, από την Αυστραλία κρέας και στη δεκαετία του 50 και του 60 η Βραζιλία 48% του, του μηνιαίου ΑΕΠ το δαπανούσε στην αγορά ακριβών προϊόντων. Σήμερα αυτοί ε, οι ίδιοι Βραζιλιάνοι μόνο το 18% του μισθού τους χρησιμοποιούν για τη διατροφή και όχι το 50% που ήταν, χρησιμοποιούσαν πριν από 40 χρόνια. Οπότε με τα υπόλοιπα χρήματα ο κάθε Βραζιλιάνος μπορεί να επενδύσει στον οικοκυριό του, στα παιδιά του, στην προσωπική του ευημερία. Η Βραζιλιάνικη Γεωργία δεν είχε μόνο οικονομικές ε, ε, οι δημοσιονομικές συνέπειες, οι συνέπειες στις εισαγωγές στην απασχόληση, στο εμπορικό ισοζύγιο. Το βασικό πλεονέκτημα της βραζιλιάνικης γεωργίας κτηνοτροφίας ήταν κοινωνικού χαρακτήρα. Αύξηση της κοινωνικής ευημερία. Γιατί τότε λάβαμε μια πολύ ευφυή πολιτική απόφαση στη δεκαετία του 60. Επιλέξαμε την αυτάρκεια, την επισητιστική μας αυτάρκεια. Γι' αυτό και στην Μπράγκο, που είναι από τις μεγαλύτερες ε, ερευνητικές εταιρείε του κόσμου και που σήμερα συνεργάζεται με πάνω πολλές χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, προσπαθήσαμε να βρούμε και να χαρακτηρίσουμε ε, τους σπόρους που εισαγάγαμε από την Ευρώπη, πώς θα τους προσαρμόσουμε στο δικό μας κλίμα και στις δικές μας καιρικέ ε, καιρικές συνθήκες. Οπότε αυτοί οι σπόροι που ήρθαν από την Ευρώπη και από άλλες περιοχές του κόσμου ήταν πολύ σημαντικές για μας γιατί έτσι καταφέραμε να αναπτύξουμε τις ειδικότητέ μας λαμβάνοντας υπόψη το τροπικό μας κλίμα και τις δικές μας καιρικέ συνθήκες. Αυτή ήταν η σημαντική επανάσταση που υλοποιήσαμε στην Βραζιλία. Μετατρέψαμε δηλαδή προϊόντα δικά σας ε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου ε, και τα προσαρμόσαμε στη δική μας ε, πραγματικότητα. Ε, η γενετική ε, των βοηδών ε, μας ήρθε από την Ινδία και έχουμε τεράστιο χρέος ευγνωμοσύνης προς την Ινδία γιατί χάρη στην γενετική κληρονομιά των βοηδών από την Ινδία αναπτύξαμε τη δική μας κτηνοτροφία και έχουμε ελεύθερους ανοιχτούς βοσκοτόπους όπου οι αγελάδες μας ε, ελεύθερα ε, ε, μπορούν να κυκλοφορούν στα μεγάλα χωράφια. Και χάρη στην τεχνολογική ανάπτυξη οι παραγωγοί επένδυσαν στο έδαφος των βοσκοτόπων ώστε οι μερικοί βοσκότοποι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δημητριακών και σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και καμία ανησυχία από το 27%, το 27, από το 27% το, της επικράτειας, 237 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή που προορίζονται στην γεωργική παραγωγή, μόνο 7 εκατομμύρια εκτάρια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζαχαροκάλαμου για την εθανόλη μας. Αν διπλασιάσουμε την έκταση αυτή, ακόμη και τότε ελάχιστη έκταση θα αφιερώσουμε στην παραγωγή της εθανόλης. Και το κέρδος για το περιβάλλον, για την κοινωνία, για τις κλιματικές αλλαγές θα είναι να αποφύγουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Και αυτό το κέρδος είναι ανεκτήμητο. Ε, στη Βραζιλία είχαμε δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Την ε, ανάπτυξη της ε, παραγωγής του ζαχαροκάλαμου και τα ποτάμια που σώσαμε και τη χρήση του ύδατος ώστε να χρησιμοποιήσουμε υδροελεκτρική ενέργεια που είναι πολύ καθαρή ενέργεια. Η υδροελεκτρική ενέργεια είναι η καθαρότερη ενέργεια που υπάρχει. Καταφέραμε χάρη στην αξιοποίηση των ποταμών μας να αυξήσουμε την υδροελεκτρική μας ενέργεια. Βλέπω εδώ τον πρόεδρο να κρατάει το σφυρί και θα προσπαθήσω να υπακούσω. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για την αποψήλωση αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί πέρυσι όλοι ε, αναγνώρισαν την προσπάθεια και τα επιτεύγματα της Βραζιλίας ό,τι αφορά τον περιορισμό της αποψήλωσης. Και στην Κοπεχάγη, στη Δανία, αναλάβαμε τη δέσμευση να μειώσουμε την αποψήλωση στη ζούγκλα του Αμαζονίου που ήταν 29 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέχρι το 2020 αναλάβαμε την δέσμευση να μειώσουμε κατά 80% αυτή την αποψήλωση και 10 χρόνια πριν το 2020 έχουμε μειώσει την αποψήλωση κατά 70% και την αποψήλωση του Αμαζονίου. Και σήμερα οι άπιστοι θωμάδες μπορούν με δορυφορικά συστήματα και με ακριβείς φωτογραφίες να ελέγξουν αν λέμε αλήθεια ή λέμε ψέματα ο διεθνής τύπος ε, ε, επένεσε τη Βραζιλία για την ε, προσπάθεια αυτή. Και σήμερα έχουμε μια τελείως διαφορετική εντύπωση και ένα διαφορετικό όραμα για τον Αμαζόνιο. Σήμερα είμαι Υπουργό Γεωργίας. Αν με ρωτούσατε πριν από μια δεκαετία τι γνώμη έχω για την ε, σημασία του Αμαζονίου. Ίσως τότε από άγνοια θα σας έλεγα ότι ο Αμαζόνιος δεν έχει καμία αξία, ότι είναι υπερβολές των οικολόγων. Σήμερα όμως ως ηγέτης της πολιτικής τάξης, ε, ε, που ήμουν 20 χρόνια σε αυτήν την πολιτική τάξη και σήμερα ως υπουργό Γεωργίας τονίζω τη σημασία που έχει η ζούγκλα του Αμαζονίου και το τροπικό δάσος. Γιατί αν θέλουμε ε, αν, λέω στους γεωργούς, ε, αν προστατεύσουμε το περιβάλλον θα προστατεύσουμε τα εισοδήματά μας, γιατί χρειαζόμαστε τη ζούγκλα του Αμαζονίου για να εξασφαλίσουμε βροχοπτώσεις στις γεωργικές μας εκτάσεις. Και φυσικά ε, ο περιβαλλοντικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και η βιοπικιλότητα που υπάρχει στον Αμαζόνιο είναι τεράστια. Δεν γνωρίζουμε το 10% αυτού του πλούτου του φυσικού που υπάρχει στον Αμαζόνιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι κλιματικές αλλαγές. Φυσικά και μα απασχολούν οι κλιματικές αλλαγές. Φέτος αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες ε, ε, στο Σαο Πάολο, στην πολιτεία Παρανά, στο νότιο της πολιτείας Μιναζεράη, στο κέντρο της πολιτείας Γκογιάς. Είχαμε προβλήματα σημαντικά λειψιδρίας σε πολλές μας πολιτείες και στα τέλη του προηγούμενου έτους και στις αρχές του τρέχοντος έτους. Σήμερα χρειαζόμαστε και αναγνωρίζουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Πολλά προβλήματα θα τα είχαμε αποφύγει αν ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι και αν είχαμε κάνει πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων μας πόρων. Κάποιοι κυβερνήτε, βέβαια δεν θέλουμε εδώ να βρούμε από διαπομπέου τράγου και να διαχωρίσουμε του φταίχτε από του αθώου. Αλλά κάναμε λάθη στι κλιματικέ αλλαγέ. Εκεί χρειαζόμασταν περισσότερη έρευνα. Ε, έπρεπε να αποφύγουμε προϊόντα που χρειάζονται περισσότερο νερό για την παραγωγή. Αν δούμε, πόσα λίτρα νερού χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν για το ρύζι, ενώ σήμερα χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερο νερό για την παραγωγή του ίδιου ρυζιού και έχουμε μειώσει περίπου κατά 70% τη χρήση του νερού ανασπόρο ρυζιού, μόνο χάρη στη χρήση της τεχνολογίας. Έχουμε το 12% των υδάτινων αποθεμάτων του πλανήτη στη Βραζιλία. Έχουμε 30 εκατομμύρια εκτάρια στη Βραζιλία που μπορούν να αρδεύονται. Από αυτά τα 30 εκατομμύρια αρδεύουμε μόνο τα 5 εκατομμύρια εκτάρια. Οπότε έχουμε ένα σημαντικό κέρδος αν αρδεύουμε σωστά με ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σημαντικό τμήμα αυτών των εκτάσεων για να αυξήσουμε την παραγωγή μας και την παραγωγικότητά μας, χωρίς να χρειαστεί να κόψουμε ούτε ένα δέντρο επιπλέον. Μόνο χρησιμοποιώντας πιο ορθολογικά τους υδάτινους πόρους, γιατί με την άρδευση μπορούμε εκεί που έχουμε δύο χωράφια να αρδεύουμε, με μια πολύ πιο ορθολογική διαχείριση μπορούμε να αρδεύουμε τρία. Μου επιτρέπετε λίγο ακόμη να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε. Okay. questão σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ηθαγενών, των αυτόχθων πληθυσμών. Ε, οι χώρες και οι Υπήροι ανακαλύφθηκαν, ε, ε, έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης, οικειοκρατίες. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μάλιστα είμαστε υπερήφανοι για την πορτογαλική απεικιοκρατία, γιατί χάρη σε αυτήν καταφέραμε στη Βραζιλία να γίνουμε ε, μια τεράστια περιοχή, μια χώρα με μία και μόνη γλώσσα. Αλλά έγινε και κάποια λάθη στη διαδικασία αυτή. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 11% της ε, βραζιλιάνικης ε, επικράτειας ή μάλλον 13% της χώρας, της επικράτειας, δηλαδή 115 εκατομμύρια εκτάρια, προορίζονται σε 816.000 ηθαγενείς. Επαναλαμβάνω. 115 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή το 13% της Βραζιλιάνικης επικράτειας, ε, ε, προορίζονται σε 816.000 Ινδιάνους, Ιθαγενείς. Δηλαδή 11% ουσιαστικά του συνόλου της, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είναι σαν να έχουμε 38, 38 ε, φορές το Βέλγιο, την έκθεση του Βελγίου. Είναι μια έκθεση που δίνεται, που ανήκει στους Ιθαγενείς της Βραζιλίας. Αν έμεναν αναπάντητα κάποια ερωτήματα, σας ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να είχα απαντήσει για το θέμα των γυναικών, των νέων, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγος. Είμαι στη διάθεσή σας να συνεχίσω, αλλά μια και εξάντλησα το χρόνο, δεν έχω καμία αντίρρηση να σας στείλω γραπτός τις απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις που σημείωσα με πολύ προσοχή και φροντίδα και στοργή. Κυρία Υπουργέ, χαιρόμαστε ιδιαίτερως ε, για αυτά που μας είπατε και είναι πολύ σημαντικό η υπουργό ε, της κυβέρνησης μιας τόσο μεγάλης χώρας, ε, μιας τόσο σημαντικής γεωργίας να έχει τέτοια αντίληψη για τόσο σημαντικά θέματα που είναι σημαντικά όχι μόνο για τη Βραζιλία αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί ε, ο φυσικός πλούτος της Βραζιλίας ε, και η γεωργία της ε, είναι τεράστια και εξίσου τεράστια είναι η ευθύνη της για τα περιβαλλοντικά θέματα και η ευθύνη της απέναντι σε επερχόμενες γενές. Και το ίδιο ισχύει και για μας και πολύ συχνά το επισημαίνουμε. Όπως είπα, η παγκοσμιοποίηση, η παγκόσμια αγορά μας υποχρεώνει να ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά κατά τη χάραξη της κοινή μας γεωρικής πολιτικής. Γιατί η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ένα άλλο επίπεδο ε, που παραγωνίζει πια τις διμερείς λύσεις. Θα πρέπει από κοινού να φτιάξουμε το μέλλον μας γιατί μόνο έτσι θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα και όχι ο καθένας μόνος του. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Λυπούμε που δεν ευχαρίστησα μεμονωμένα το κάθε μέλος της αντιπροσωπείας σας. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία που είχαμε να ανταλλάξουμε απόψη και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μην ξεχνάτε ότι οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου αντιπροσωπεύουν 28 διαφορετικές χώρες. Και μάλιστα αυτή η συνεργασία και αυτή η συζήτηση έχει ιδιαίτερο βάρος και σημασία. Σας ευχαριστώ και προσβλέπουμε σε θετικές εξελίξεις. Ευχόμαστε καλή τύχη για αυτή την τεράστια χώρα που είναι η Βραζιλία, για τους κατοίκους της, για τους γεωργούς τους και για τις τεράστιες προκλήσεις που έχει να σητήσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτού του σημείου και χαρήκαμε ιδιαίτερως ε, για την ευκαιρία που είχαμε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι το θέμα της, ε, είναι το θέμα της ε, βιολογικής γεωργίας. Η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Χόισλινγκ. Του φάγαμε λίγο χρόνο, ελπίζω να μας συγχωρέσει γιατί ήταν πολύ σημαντικό το προηγούμενο θέμα. Σας αποχαιρετώ λοιπόν κύριε Υπουργέ, ευχαριστώντας σας και πάλι θερμά για την ε, επίσκεψή σας. Θα ήθελα να ξεπροβοδίσω την ε, Υπουργό, δίνοντας το λόγο στον κύριο Χόισλινγκ για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από μένα ο κύριος Χόισλινγκ στην παρουσίαση της έκθεσής του. Κύριε Χόισλινγκ, τι γίνεται. Περιμένουμε την παρουσίασή σας, κύριε Χόισλινγκ. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ. Προσπαθώ να ξεκινήσω, για να μην χάσουμε και πολύ χρόνο. για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαρτίου 2014 για μια νέα ε, τροποποίηση του κανονισμού ΙΚΟ. Δεν ήταν ε, και ενθουσιώδης η αντίδραση από πλευρά του Κοινοβουλίου στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να το πω ήπια. Κατέθεσα την έκθεσή μου 300 53 συντροπολογίε που κατατέθηκαν στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό καταδεικνύει το βαθμό τη ε, τροποποίηση που επιθυμούμε. Ελπίζουμε και για το καλά του κλάδου αλλά και για την ε, προστασία των καταναλωτών να ρυθμίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό. Ένα στοιχείο ήθελα να τονίσω εξ αρχή, ο μεγάλο αριθμό πράξεων κατά ταξιοδότηση. Προσπαθήσαμε στο βαθμό του δυνατόν να τι περιορίσουμε. επαναφέροντας σε πολλές περιπτώσεις τον παλιό κανονισμό. Δεν είναι δυνατόν. Μία νέα τέτοια νομοθετική πρόταση να την φορτώσουμε με τόσες νομικές αβεβαιότητες, όπου και στη συνόχεια να δίνουμε λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μελλοντική διαμόρφωση του κανονισμού. Εγώ υποστηρίζω την νομική ασφάλεια για όλο τον κλάδο. Και έτσι λοιπόν ε, να υπάρχουν λιγότερες ε, πράξεις κατά ταξινοδότηση. Ένα θέμα που προκάλεσε έντονες συζητήσεις ε, στα πλαίσια του κλάδου, αλλά και μεταξύ κρατών μελών, είναι το θέμα του κατά πόσον θα εισαχθούν νέες οριακές τιμές για οικολογικά προϊόντα. Μηδενική δηλαδή ανοχή για τα φυτοφάρμακα. Εγώ είμαι ξεκάθαρα κατά. Είμαι ρητά κατά της πρότασή αυτής γιατί πιστεύω ότι αυτό θα καταπίεζε την αρχή της, ε, του υπεύθυνου. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε αυτό να μείνει στα χέρια της ε, ρύθμισης από τον τομέα των οικολογικών προϊόντων. Είτε θα πρέπει να ισχύουν αυτές οι ωραίες τιμές για όλους, είτε όχι. Και να μην υπάρχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα να μην ε, κάνουμε τη συζήτηση λοιπόν αυτή για τις οριακές τιμές που αποτελεί και ένα οριακό, ένα μικρό πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα του έλεγχου της διαδικασίας. Γιατί η, βιολογική παραγωγή ξεκινάει από την παραγωγή του και από το έδαφος. Δεν περιλαμβάνει μόνο τα φυτοφάρμακα. Θα ήταν πολύ μεγάλος περιορισμός το να το περιορίσουμε αυτό μόνο σε θέματα χρήσης μη φυτοφαρμάκων. Ως εκ τούτου, θέλουμε να τεθεί και το θέμα της ευθύνη του παραγωγού, να ενισχυθεί η ευθύνη του παραγωγού. Θα πρέπει να αναφέρουν ε, περιπτώσεις μόλυνσης, θα πρέπει να παρεμβαίνουν τα κράτη-μέλη και ως εκ τούτου η, προστασία του καταναλωτή αποτελεί ανώτερο αγαθό. Συμφωνώ. Αλλά αυτό αφορά και τους ελέγχους οι οποίοι θα πρέπει να υπάρχουν. Πιστεύω, και αυτό κατέστη σαφέ ε, στην επεξεργασία του κειμένου, σε όλη τη διαδικασία, ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο και ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο ο παλιό κανονισμό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι πολύ διαφορετικά τα συστήματα ελέγχου, είναι πολύ διαφορετικέ οι ερμηνείε του πότε πρέπει να αποσυρθεί και πότε όχι ένα προϊόν και δεν έχουμε βάσεις δεδομένων εκτενής. Δεν είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει πού χρησιμοποιούνται οικολογικοί σπόροι, βιολογικοί σπόροι και πού όχι και σε τι βαθμό. Εγώ λοιπόν ζητώ την υποστήριξή σας προκειμένου όπως και σε άλλους τομείς να υπάρχει μια υπηρεσία για την βιολογική παραγωγή, να εναρμονιστούν τα συστήματα στην Ευρώπη προκειμένου να προχωρήσει πολύ περαιτέρω ο κλάδος και στις εισαγωγές που αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα να υπάρξει εναρμόνιση. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε να υπάρχουν τόσο πολλά διαφορετικά συστήματα για τον έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε το τι ακριβώς γίνεται και πιστεύω ότι με μια τέτοια υπηρεσία βιολογική, βιολογικής παραγωγής θα πετύχουμε την εφαρμογή των ίδιων προτύπων προκειμένου να εναρμονιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι ένα στόχο ο οποίο έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις βιολογικούς σπόρους, τη βιολογική εκτροφή ζώων, συμφωνώ. Αλλά ναι, μην υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα. Θα πρέπει στους βιολογικούς καλλιεργητές και παραγωγούς και εκτροφής να δώσουμε την ευκαιρία και πιστεύω ότι με ένα νέο κανονισμό θα πρέπει να πετύχουμε στην Ευρώπη την πραγωγή των ε, προτύπων αυτών. Αλλά προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και στις, ε, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κάθε, του κάθε κράτους μέλους. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το στόχο, συμφωνούμε. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στον τρόπο επιτεύξης του στόχου αυτού. Αν μια περιοχή, για παράδειγμα, έχει λίγου ε, βιολογικούς εκτροφεί, προφανώς δεν θα αγοράζει και πολλές βιολογικές ε, τροφές, ε, ζωοτροφές. Και θα πρέπει να βρούμε ευέλικτου κανόνες για την εφαρμογή και τη μεταστροφή σε βιολογικούς τρόπους καλλιέργεια. Ένα θέμα το οποίο έθεσα ακόμα και το συζητήσε και ο κλάδο πολύ και πιστεύω ότι και για μα είναι σημαντικό κατά πόσον θέτουμε πρότυπα σε ό,τι αφορά την εκτροφή των ζώων. Εγώ δύο σημεία ανέφερα, όπου πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά τους βιολογικούς εκτροφείς. Τρεις ε, χιλιάδες τόνοι νομίζω ότι είναι επαρκής, θα πρέπει να πούμε. Συγγνώμη, όταν μιλάμε για τον αριθμό των ζώων. Τα όρια αυτά μπορεί να συζητηθούν. Σε ό,τι αφορά ε, τα πτηνά, τις ε, αγελάδες. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει αυτό μια βάση για συζήτηση. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το θέμα των ελέγχων. Το θέσαμε και αυτής εξ αρχής, Είμαι κατά της αντικατάστασης των αιτήσεων ελέγχων από ελέγχους κινδύνου. Πρέπει να συνεχιστούν γιατί έχουν την εμπιστοσύνη των γεωργών και των εκτροφέων για τη αυτή έλεγχη. Αυτό με τη σειρά του δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποστρεχθεί το σύστημα με ελέγχους κινδύνου. Άρα το να στηριχτούμε μόνο σε αυτή την ανάλυση κινδύνου πιστεύω ότι δεν επαρκεί. Θα πρέπει να μεταρρυθούν και αυτοί οι ετήσιοι έλεγχη. Πιστεύω ότι το σύστημα των ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής έχει αποδείξει την αξία του. Και θα πρέπει λοιπόν να το κρατήσουμε και να το βελτιώσουμε περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά τους βιολογικούς ελέγχους, πιστεύω ότι θα πρέπει να θρηχθούμε σε, βιολογική, σε ε, περιφερειακά πρότυπα. και πιστεύω ότι να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός, μια ευρωπαϊκή ρύθμιση δεν θα, έχει, δεν θα αποφέρει καρπούς. Δεν θέλω να σας εξηγήσω και να σας παρουσιάσω και τις 352 τροπολογίες. Έχουν μεταφραστεί στις πιο πολλές γλώσσες. Κάποιες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στις πολυάριθμες τεχνικές συζητήσεις και τους κοιόδες συζητητές να ευχαριστήσω για τις συζητήσεις ε, πριν από την ανάλυση της πρωτοβουλίας και για τις επικοδομητικές ε, ανταλλαγές απόψεων. Ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία φέτος, γιατί αυτό το επιθυμεί διακάως ο κλάδος, να υπάρξει επιτέλους σαφήνεια σε ό,τι αφορά την ε, προώθηση της οικολογικής παραγωγής και εκτροφής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ. Θα συνεχιστεί φυσικά η συζήτηση, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι μεταφράσεις. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει προθεσμία για την ε, κατάθεση τροπολογιών τη 12η Ιουνίου. Μην ξεχνάτε ότι στις 5.30 θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα του κυρίου Χόισλινγκ. Παρακαλώ συλλάβουν το λόγο να μην ξεπεράσουν το ένα λεπτό για να προλάβουμε να πάμε εγκαίρως στην κοινή συνεδρίαση. Ο κύριος Ρίνς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτάκι είπαμε. Jetzt klappt. Ich glaube, er sieht mich immer noch nicht. Herr Vorsitzender, vielen, vielen Dank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 Έχετε δίκιο ότι κρίμα είναι που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για την ουσία της συζήτησης. Ο κύριος Αντριέ. Ε, oui, merci, Monsieur le είναι παράλογο να έχουμε μια τέτοια προθεσμία για τις τροπολογίες για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Λυπάμαι γι' αυτό και μάλιστα να γίνεται μια ζώρικα βιαστική συζήτηση μέσα σε 32 λεπτά. Γιατί τα θέματα που έθεσε ο Μάρτιν είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεν έχει νόημα μέσα στο λεπτό να πω τίποτα. Να χαιρετήσω όμως την τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε ο Μάρτιν. Αναφέρθηκε σε 350 τροπολογίες Νομίζω ότι αναζητούμε όλοι μια γεωργία πραγματικά ευρωπαϊκή με ένα πεδίο εφαρμογής των κανονισμών του μικτού χαρακτήρα της πολιτικής με άλλες πολιτικές, της συνεργασίας, του συντονισμού, ιδιαίτερα σε το ΜΙΣΟ όπως η διασταυρώση ειδών η έρευνα στη γενετική και για τα φυτικά προϊόντα και για τα ζωικά προϊόντα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει για την έκθεση αυτή μια πραγματική συζήτηση έτσι ώστε να εξετάσουμε σοβαρά τις προτάσεις του εισηγητή. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Χάουσλινγκ για την διαθεσιμότητά του και την ιδιαίτερα συνθετική δουλειά την οποία πέτυχε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να πω ότι για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό αποτελεσματικά θα πρέπει να έχουμε μία μακροπρόθεσμη αντίληψη. Ε, βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος τομέας η γενετική βιολογία είναι ένας τομέας ιδιαίτερα πλούσιος αλλά ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα παραδοσιακά στοιχεία της παραγωγής. Τα διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να μας επιτρέψουν να αναφερθούμε και στην εξωτερική αυτή υπηρεσία, η οποία μου δημιουργεί κάποια θέματα, όχι μόνο για θέματα κόστους, αλλά για τη θεωρή τον βιολογικό τομέα σαν ένα τομέα άλωση, προς άλωση, προς εκμετάλλευση και όχι τόσο ε, σαν κάτι το φυσιολογικό. Θα πρέπει λοιπόν η μεταβατική περίοδος αυτή να είναι πραγματικά μεταβατική και όχι κάτι το απόλυτα δεσμευτικό για το μέλλον. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μετά την υποβολή των τροπολογιών θα έχουμε εκτενή συζήτηση για την εξέταση των τροπολογιών. Δεν είναι η τελευταία φορά που συζητούμε αυτό το θέμα. Η κυρία Μίλλερ. Ναι, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματο ε, του σκιώδου εισηγητή μα, ο οποίο είναι δυστυχώ ακόμα στο αεροδρόμιο. Καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή και την ε, ισορροπή έκθεση του κυρίου Χόισλικ. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ε, ρεαλιστική προσέγγιση την οποία διαπιστώνουμε στην έκθεση και στην βασική νομοθετική πράξη, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν τα στοιχεία αυτή. αυτά. Λέμε σαφέστατα όχι στις οριακές τιμές αυτές. Η αρχή του παραγωγού σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του κόστους μέχρι 5.000 ευρώ Ανά έτος πιστεύουμε ότι είναι πολύ ψηλό το πόσο αυτό το θέμα της οικολογικής υπηρεσίας μπορούμε να το συζητήσουμε ή το εμπόριο με τις τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι οι προτάσεις που κάνετε εδώ είναι σημαντικές, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε άκρη μετά τα όρια στο θέμα της εκτροφής Θα πρέπει να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό και σε γενικές γραμμές είμαστε πραγματικά θετικά έκπληκτοι πρέπει να πω, από το σχέδιο πρότασης. Κυρία Χαϊτοβά. Sorry, sorry, Chair. Thank you, Chair. First of all... Συγγνώμη, Πρόεδρε, και σας ε, ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, κύριε Χόισλινγκ, για την πολύ καλή δουλειά. Προσωπικά δεν, πιστε... δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε το νέο κανονισμό. Πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε μεγάλη γραφειοκρατία. Να εκφράσω την ανησυχία μου για κάποια βασικά θέματα. Η παραλληλή παραγωγή αναφερθήκατε στα θέματα αυτά, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να δοθεί χώρος στους παραγωγούς για να έχουν και παραδοσιακή και βιολογική καλλιέργεια. Η Επιτροπή προτείνει μία ένα σύστημα ελέγχων βάσει κινδύνου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και το κόστος. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εξαίρεση από τις πιστοποίησεις μόνο για προσυσκευασμένα προϊόντα. Προτείνει ο εισηγητής. Αυτό μα περιορίζει πολύ, πιστεύω, σε σχέση με τον τρέχοντα κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ στη σημερινή συζήτηση, αλλά στις συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα. Και είναι παράλογο να μην έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας για να μιλήσουμε για κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να το λάβει υπόψη αυτό η γραμματεία, να έχουμε για κάθε συζήτηση τρίλεπτη δυνατότητα ομιλίας πρέπει να μελετήσουν αυτή την πρόταση, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην Ολομέλεια, δεν μπορούμε να, να μιλήσουμε και σε επιτροπή, τότε τι κάνουμε εδώ πέρα. Προέρχομαι λοιπόν από μια χώρα η οποία έχει υψηλή παραγωγή βιολογικών γεωργικών προϊόντων και γι' αυτό θα καταθέσω αρκετές τροπολογίες και υπάρχουν θέματα συγκεκριμένα όπως το θέμα της πορείας σαν παράδειγμα είναι θέματα στα οποία θα καταθέσω όπως είπα αρκετέ τροπολογίες και σας παρακαλώ να ανταρρυθμίσετε έτσι τα πράγματα έτσι ώστε για ένα τρίλεπτο να μπορούμε να πάρουμε το λόγο. Όντως, μπορούμε να προβλέψουμε και δεύτερη συζήτηση για να έχουμε τη δυνατότητα για πιο εκτενείς παρεμβάσεις. Αλλά σήμερα έγινε μια ενημέρωση για αυτό το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Μετά την υποβολή τροπολογιών θα γίνει νέα συζήτηση. Κύριε Κέστιγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Χόισλινγκ, τον εισηγητή. Ένας ε, πράσινος ε, ζητά ανώτατες τιμές ε, και τέτοια συστήματα, τι τι να πω, ε, αστείο. Αλλά πέρα από αυτά, να σας πω για τα βιολογικούς σπόρους και τις βιολογικές τροφές. Θα ήθελα να υπάρχουν κίνητρα. 85% των σπόρων είναι στο, στα χέρια τριών ομίλων από ό,τι φαίνεται στην Ευρώπη. Δεν μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί η αγορά σπόρων θα πρέπει να δοθούν πραγματικά κίνητρα για να υπάρχει εξέλιξη και για τους παραγωγούς ευρωπαϊκών σπόρων. Χρειαζόμαστε επίσης εκμεταλλεύσεις, ε, εξαιρέσεις για τις εκμεταλλεύσεις στις ορεινές περιοχές. Και εδώ οι βιολογικές καλλιέργειες αποτελούν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να υπάρχει μέλλον για τις εκμεταλλεύσεις αυτές. Αυτό που δεν κατάλαβα λόγω της, ε, του μεγέθους των εκμεταλλεύσαν, αλλά αυτό δεν αφορά άμεσα την Αυστρία. Γιατί, τι διαφορά έχει το να έχουμε 2.999 χείρους ή 3.001. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα δεν υπάρχει διαφορά. Έχει να κάνει αυτό με την μέθοδο εκτροφής. Αλλά αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να το συζητήσουμε πέραστατα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόταση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτείται περισσότερος χρόνος και ζητώ από τον Πρόεδρο και από την Γραμματεία να ρυθμίσουν τα πράγματα καλύτερα. Και εγώ είμαι Ισπανίδα, έχουμε πολύ υψηλή παραγωγή οργανικών προϊόντων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα μέτρα έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο θα συμβιώσει η βιολογική παραγωγή με την παραδοσιακή, τη συμβατική καλύτερα παραγωγή. Πρέπει να καταστήσουμε αυτή τη συμβίωση εφικτή. Θα δεχθούμε λοιπόν τις προτάσεις αλλά με κάποιες τροπολογίες. και υπάρχουν πολλά τα οποία θα πρέπει να πούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον βασικό κανονισμό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης το άρθρο 20. Νομίζω ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει σήμερα είναι πάρα πολύ αρνητική. Και εδώ θα υπάρξει μια τροπολογία νομίζω σημαντική. Υπάρχει επίσης και το θέμα με την no confundan comprendo que usted es verde y comprendo su ideología pero a veces Εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να γίνει στον τομέα της παραγωγής, ε, της κτηνοτροφίας ε, ε, και της οργανικής παραγωγής. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να θέσω το θέμα της διαχείρισης του χρόνου. Δύο ώρες σχεδόν αφιερώσαμε ε, στη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν λέω, τη γεωργία τη Βραζιλία, αλλά για ένα σημαντικό θέμα όπου έχουμε το καθεστώ του συνομοθέτη, ε, έχουμε 15 λεπτά. Πιστεύω ότι κάπου κάτι δεν πάει καλά. Ένα θέμα θα αναφέρω, το θέμα των οριακών τιμών σε μια χώρα όπως την Ιταλία για παράδειγμα, όπου το θέμα των οριακών τιμών οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα γιατί τα θέματα μόλυνσης των συμβατικών ε, καλλιεργειών σε βιολογικές ε, καλλιέργειες είναι σημαντικό. Και κάποιες, ε, πολλές βιολογικές εκμεταλλεύσεις αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον βιολογικό τρόπο παραγωγής λόγω των οριακών τιμών αυτών. Αν είναι έτσι, μπορούμε να καταργήσουμε την βιολογική παραγωγή. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τι εμπειρίε τη Ιταλία και να καταπιστώσουμε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω έχει, μάλλον δεν βγάζει νόημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χόισλινγκ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. η βιολογική παραγωγή στην ε, Βουλγαρία ε, κάπως αντίστροφη. Στο 196 μιλούμε τον έλεγχο της ε, παρατυποποίησης των βιολογικών προϊόντων. Το σημείο 3, το 3 μιλά για, έλεγχο, για μελέτη επιπτώσεων. Πιστεύω ότι για να διαφυλάξουμε την καθαρότητα της βιολογικής παραγωγής θα πρέπει τους ελέγχους να τους κρατήσουμε ετησίως για όλους τους παραγωγούς γιατί αυτή είναι μια εγγύηση ποιότητας της βιολογικής μας παραγωγής. Δεν θα πρέπει να καταργήσουμε τέτοιους ελέγχους. Επίσης, το 345 λέμε ότι τα κριτήρια θα θεσπιστούν αργότερα. Τι εννοείται, κύριε Χόισλινγκ? Πότε δηλαδή θα οριστούν τα κριτήρια? Οι ομαδικές πιστοποίησεις, κάτι καινούργιο που θα μειώσει το γραφειοκρατικό άχθος. Οι παραγωγοί όμως πρέπει να ξέρουν τις συνθήκες και τους όρους που θα πρέπει να πληρούν. Η, βιολογική, η παραγωγή βιολογικής γεωργίας μου τηλεφώνησαν ανίσχυοι και είπαν ότι σε αυτές οι ομαδικές αιτήσει για προτυποποίηση αποβούν εις βάρος της ποιότητας των βιολογικών προϊόντων. Επίσης, τι γίνεται με τις ποικιλίε και τα διάφορα είδη σπόρων. Για παράδειγμα, ποικιλίε ε, φρούτων και λαχανικών. Πολύ σημαντικό θέμα οι ποικιλίε. Γιατί μπορούμε να έχουμε μια ποικιλία που να ευδοκιμεί ιδιαίτερα σε μια περιοχή και έτσι να διατίθεται στην αγορά. Και έτσι μπορούμε ταυτόχρονα να προωθούμε την τοπική παραγωγή ενισχύοντας και την καινοτομία στον τομέα. Θα σας υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χάουσλινγκ. Είμαι παλαιό μέλος, αλλά έλειπα γιατί ε, τώρα ήρθα πλέον στη θέση του Όλη Ρεν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν σε σχέση με την πρόταση αυτή, όπως η εξωτερική υπηρεσία. Σαν νομοθέτες θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε καλύτερη αλλά και λιγότερη ε, νομοθετική δραστηριότητα. Και νομίζω ότι η υπηρεσία αυτή ε, δεν έχει να προσθέσει πάρα πολλά. Τα τεστ για την αξιολόγηση των κινδύνων μπορεί ήδη να γίνουν από τις υπάρχουσες δομές και νομίζω ότι αυτή η έλεγχοι έτσι όπως προβλέπονται είναι απολύτως επαρκείς. Απαιτείται να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, να υπάρχει περισσότερη λογική στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας για να βελτιώσουμε την παραγωγή. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες. Σας ευχαριστώ. Ε, μέχρι τη στιγμή που έγινε η πρόταση αυτή, η περισσότερη παραγωγή οργανικών προϊόντων μας, ε, μας συμπαθούσαν. Αλλά η πρόταση αυτή αλλάζει τις απόψεις τους. Θα είναι αδύνατον στη χώρα μου κάτω από τους κανόνες αυτούς να καλλιεργεί ε, κανείς οργανικά προϊόντα. Είναι περίπλοκο, η αγορά είναι ευαίσθητη και εύθραυστη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εδώ είναι ότι εμείς ελέγχουμε καλά την παραγωγή οργανικών προϊόντων μέσω του Soil Association. Αλλά από ό,τι φαίνεται η πρόταση αυτή λέει ότι η παραγωγή οργανικών προϊόντων είναι καλύτερη από οτιδήποτε άλλο και δεν θα πρέπει να επιμολυνθεί από οποιαδήποτε άλλη μορφή πορείας. Λοιπόν, ξέρετε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στους οποίους υπάρχουν ε, ε, μίξεις και επιμολύνσεις και σε σχέση με τα περιτώματα των πτηνών και σε σχέση με άλλα είδη τα οποία στη συγκεκριμένη προϊόντα τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε ακόμα εξετάσει. Ο κύριος Φεντερέι αν δεν θέλει ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Φέγο. Ε, εδώ παρακαθήμενος ε, με μπέρδεψε. Με ικανοποίηση διαβάσαμε την έκθεση του κυρίου Χόισλινγκ που ε, μιλάει ιδιαίτερα για την εδαφική ταυτότητα των βιολογικών προϊόντων και την απόρριά της, δηλαδή την πρόθεση ε, βροχαίων κυκλωμάτων και πρόθεση των τοπικών προϊόντων. Όλα αυτά είναι καλά και άγια, απαραίτητα. Να σταθώ σε ένα σημείο που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που μας ε, ε λυπεί στην πρότασή του είναι ότι δεν χτυπά το κοινωνικό ντάμπινγκ, γιατί σε ορισμένες περιοχές η βιολογική γεωργία ε, βρίσκεται δυστυχώς ε, σήμερα ε, στην παγίδα των πολύ ακριβών προϊόντων με υπερβολικό κόστος παραγωγής. Θα πρέπει το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ να ληφθεί υπόψη και στη μελέτη αυτή για τη βιολογική γεωργία. Γιατί ε, η πρόσληψη φθηνού εργατικού δυναμικού 10 ευρώ την ώρα εμποδίζει την υλοποίηση του στόχου προώθησης ε, των βιολογικών προϊόντων χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ευχαριστώ τώρα κύριο Φέντερλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας τη σημασία του να υπάρχει η ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή γιατί για μας ως μέλη είναι πάρα πολύ υποφελές για να καταλάβουμε τι ακριβώς ε, έχει σημασία για τον κάθε και προκειμένου να έχουμε την ε, σωστή αντιμετώπιση όταν θα γίνει η ψηφοφορία. Ο εισηγητής κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία που θα πρέπει να καλυφθούν. Τρία συγκεκριμένα. Το θέμα του κατά πόσον μπορεί να υπάρχει παραγωγή γάλακτος ή βόη κρέατος με βιολογικό τρόπο παραγωγή στο μέλλον. Στις μικτές, στα μεικτά αγροκτήματα στην Σουηδία βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατανομή του κινδύνου σε ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση της ε, βιολογικής παραγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εντάλλως πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν βιολογικές ε, μονάδες. Τώρα, για την ε, υπηρεσία βιολογικής παραγωγής, όπως είπε και ο φιλανδός συνάδελφος, δεν πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό ιδέα. Δεν θα πρέπει να υπάρξει γραφειοκρατία, να μην υπονομεύσουν με την αναπτυσσόμενη αγορά, απλά να την δώσουμε κίνητρα. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πολύ. Και να συγχαρώ τον ε, κύριο Χόισλεν για τη δουλειά που έκανε να συμφωνήσω ότι θέλουμε πιο πολύ χρόνο να καταθέσουμε τροπολογίες δεδομένου του βαθμού λεπτομέρειας. Αν τώρα, ε, για αυτούς που θέλουν να μιλήσουν πιο πολύ εδώ, μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινάμε τις συνεδριάσεις στην ώρα μας, γιατί εγώ έρχομαι εδώ κάποιες φορές και αναρωτιέμαι ειλικρινά. Είναι δυνατόν να περιμένω ο κόσμος να κάθεται και να χαζεύει και να έρχεται μισή ώρα μετά την ε, υποτιθέμενη ώρα έναρξης ε, πρόεδρε, πραγματικά σας θαυμάζω για το έργο σας. Προσπαθείτε να μαζέψετε όλα τα και να ξεκινήσουν τη δουλειά τους. Εγώ ήμουν σε, ε, σε σχολείο δουλεύα και πραγματικά όλοι ξεκινούσαμε ε, στην ώρα μας. Τι να σας πω. αν είχαμε ξεκινήσει στην ώρα μας θα είχαμε 28 λεπτά παραπάνω να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Θα λάβω υπόψη το σχόλιο σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ε, κυρία Μονίκ Παλιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χάουσλινγκ για την πρόταση του. Είναι σημαντική πρόταση και την περιμέναμε με ανυπομονησία. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τώρα λίγο τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή παρουσίασε τη συγκεκριμένη πρόταση. Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής παραγωγής είναι μεγάλη. Ένας τομέας ο οποίος από περιθωριακό έχει αρχίσει και γίνεται σφαιρικός και καθοριστικός και αποκτά μια τεράστια σημασία στην καθημερινή παραγωγή. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η παραγωγή αυτή καλύπτεται περισσότερο από εισαγωγές και όχι τόσο της αύξησης της βιολογικής παραγωγής στο εσωτερικό της Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε ανάγκη να διευκολύνουμε την είσοδο νέων γεωργών στον τομέα αυτό, ο οποίος όπως είπα αναπτύσσεται. Τρίτο στοιχείο είναι ότι το σύστημα ελέγχου δεν είναι αρκετά αυστηρό, έχει υποστεί αυστηρή κριτική από το ελεγκτικό συνέδριο και πάρα πολλά μένει να γίνουν. Τέταρτον, το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί σήμερα δεν έχει στο ίδιο επίπεδο ε, δικαιοσύνης αν θέλετε τους Ευρωπαίους παραγωγούς με τους παραγωγούς της Ευρώπης. Στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τους κανόνες έτσι ώστε τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες να υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι ότι ο Ευρωπαίος παραγωγός δεν είναι υποχρεωμένος να αγοράζει τέτοια προϊόντα. Το κάνει όμως γιατί έχει εμπιστοσύνη σε μια ετικέτα η οποία ε, δίδει για σεβασμό των κανόνων και είναι ελεύθερο εντομοκτώνων και άλλων μη επιτροπωμένων ουσιών. Αλλιώς ε, οι καταναλωτές δεν θα ε, έχουν κανένα λόγο να αγοράζουν τα προϊόντα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν τεκμηριώνεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να πω ότι σε σχέση με ένα άλλο σημείο για τα υπόλοιπα, που, τις ε, ουσίες οι οποίες παραμένουν σε ένα προϊόν και για τα ανώτατα όρια παρουσίας εντομοκτώνων και άλλων χημικών. Ακόμα και αν διασφαλίσουμε εμείς ένα σύστημα ελέγχου των προϊόντων ε, για τις απαγορευμένες ουσίες και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μπορεί να παραμένουν τέτοιου είδους ουσίες παρά τον σεβασμό των κανόνων από πλευράς των γεωργών. Και γι' αυτό λοιπόν η παρουσία αυτών των ουσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της Ένωσης, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν οι καταναλωτές να έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα προϊόντα αυτά με εμπιστοσύνη. Τώρα για τις θέσεις της Επιτροπής βλέπω ότι ο Πρόεδρος έχει το σφύρι στο χέρι. Είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής σας. Ο Επίτροπος ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του απέδειξε την δεκτικότητά του και την ευελιξία του. έτσι ώστε να εξετάζεται με σωστό και επικοδομητικό τρόπο κάθε πρόταση σε συνεργασία με τα άλλα δύο όργανα. Έτσι θα επιτρέψουμε την ανάπτυξη του τομέα αυτού. Σας ευχαριστώ κύριος Χόισλιν και πάλι ο εισηγητής μας και να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει στις 12 Ιουνίου. Επίσης με κατά την εξέταση των τροπολογιών θα διεξαχθεί και συζήτηση. Και παρακαλώ κύριε Χόισλινγκ, μπορείτε να μας κάνετε μια σύνοψη των μελλοντικών ε, συναντήσεων για να μπορούμε και εμείς να κατατοπιστούμε καλύτερα γιατί το τι μέλη ό,τι αφορά την περαιτέρω διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Επαναλαμβάνω στις 5.30 ε, πρέπει να πάμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αύριο έχουμε ελεύθερη μέρα και πέμπτη πρωί θα ψηφίσουμε. Νομίζω ότι ανέφερα τα πιο σημαντικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ για τις σύντομες προτάσεις που μου κάνατε. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να ξαναγίνει συζήτηση μετά από την κριτική που ακούσαμε και από τους συναδέλφους, γιατί όντως πολλά ζητήματα για τις βιολογικές ε, επιχειρήσεις ε, θα καθορίσουν το μέλλον τους. Πριν από το διάλειμμα το θερινό. Θα πρέπει να υπάρξει συνένεση της ε, Επιτροπής της γεωργικών υποθέσεων. Νομίζω ότι κάναμε μια συμβαστική πρόταση σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, τα χρονικά όρια. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη συζητήσει και στα κρατημέλη και μπορούμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό. Έχουμε πολιτισμικές διαφορέ μεταξύ κρατών μελών στην ε, Γερμανία, στην Αυστρία το θέμα της ε, κατανομής των επιχειρήσεων δεν είναι σημαντικό. Σε άλλες ε, χώρες, ναι, αυτό αφορά 40% των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να μην χάσουμε τις βιολογικές ε, επιχειρήσεις. Θα πρέπει σε τελική ανάλυση με τον νέο κανονισμό να αυξηθούν οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις, όχι να μειωθούν. Γι' αυτό να δούμε λοιπόν το θέμα αυτό των οριακών τιμών. Δεν θέλουμε δεν θέλουν. Οι καταναλωτέ να υπάρχουν περιορισμοί, αλλά δεν θέλουν να υπάρχουν και επιβλαβείς ουσίες. Δεν έχει νόημα λοιπόν να χρησιμοποιούμε το επιχείρημα αυτό της ασφάλειας του καταναλωτή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση, αλλά σε καμία περίπτωση, το λέω αυτό ξεκάθαρα, δεν θέλω περαιτέρω επιβαρύνσει για τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει. Θέλουμε πιο πολλέ βιολογικέ επιχειρήσει και όχι λιγότερε. Χωρίς μικρόφωνο, πρόεδρος, δυστυχώς. Επαναλαμβάνω, σε 9 θα ψηφίσουμε την Πέμπτη, να μην ξεχάσετε τις κάρτες σας και μετά έχουμε τη συνάντηση με τον αρμόδιο Επιτρόπο Χόγκαν. Τώρα μετακομίζουμε στην αίθουσα 4Q2 του Γιώζεφ Άνταλ, όπου θα συζητήσουμε το θέμα της κλωνοποίησης. Καλό απόγευμα.